I think we can start. Λοιπόν, νομίζω ότι μπορούμε να αρχίζουμε σιγά σιγά. Λοιπόν, αξιότιμοι κυρίε και κύριοι, αγαπητοί συνάδελφοι, σα καλωσορίζω θερμά στη σημερινή μας συνεδρίαση έχει διανεμηθεί η μερίσια διάταξη, το σχέδιο αυτή, αν δεν έχετε αντιρρήσει. μπορεί να θεωρηθεί ότι εγκρίνεται. Δεν διαφωνεί κανεί, οπότε εγκρίνεται η μερίσια διάταξη. Σημείο 2. Συστάσεις προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σχετικά με τις διαπραγματεύσεις για το TTIP. Ο εισηγητή μα είναι ο κ. Βιμ Βάντεν Κάμπ του ΕΛΚ είναι σημαντική αυτή η γνωμοδότηση προς την Επιτροπή Εξωτερικού Εμπορίου Διεθνούς μάλλον για να δούμε ε, πόση μεγάλη σημασία έχει ο τομέας των μεταφορών στα διατλαντικά ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά τους περιορισμούς της ε, επενδύσεις και στο καμπετά από πλευράς ΗΠΑ αλλά και θέματα ασφάλειας και κανονισμών ε, από δική μα πλευρά, 76 δοπολογίες είναι σημαντική η εναερία κυκλοφορία αλλά και η θαλάσσια. Πήγαμε στι Ηνωμένε Πολιτείε, συζητήσαμε εκεί και για το TTIP. Τα πράγματα δεν είναι πάρα πολύ απλά. Ε, περιμένω να δούμε μεγάλο ενδιαφέρον τι συνέχεια θα δώσουμε και θα δώσουμε στο λόγο στον εισηγητή τον κύριο Βίμ Κύριε Πρόεδρε, σας ευχαριστώ πολύ. Καλό μεσημέρι σε όλους σας. Καταρχάς θα ήθελα να απευθυνθώ στους συναδέλφους και ηγητές και να τους ευχαριστήσω θερμά για την ε, κριτική ε, βοήθεια ε, προβληματισμό που είχαμε από κοινού κατάληξαμε σε 76 τροπολογίες την περασμένη εβδομάδα την Τετάρτη το μεσημέρι στο Στρασβούργο συγκεκριμένα κάναμε ε, ε, μια συνεδρίαση των σκιωδών με απαρτία, παρόντες όλοι από όλες τις πολιτικές ομάδες με εξαίρεση τους μη εγγεγραμμένους και εκεί είχαμε ένα πρώτο γύρο συζητήσεων επί της ουσίας για ενδεχόμενες συμβιβαστικές ε, τροπολογίες. Και τα νέα κείμενα των συμβαστικών τροπολογιών τα έχουμε στείλει σήμερα το πρωί ότι είναι υπογραμμισμένο είναι οι συμβαστικές τροπολογίες τις οποίες συμφωνήσαμε την Τετάρτη, όπως σας είπα, στο Στρασβούργο το μεσημέρι. Δύο είναι τα προβλήματα τώρα σε αυτή την ιστορία. Πρώτον, το ζήτημα κάποιων συναδέλφων που θέλουν όλα τα θέματα TTIP να μπουν τώρα στη δική μας νομοδότηση της Επιτροπής Μεταφορών. Εγώ δεν συμφωνώ. Έχω δυσκολίες. Υπάρχει το μεγάλο ψήφισμα του Μπεντ Λάγκε. Εκεί θα μπουν τα γενικά, οι προδιαγραφές και ό,τι άλλο θέλει κανείς για το TTIP. Και δεν είναι τα θέματα των μεταφορών ε, που πρέπει να τα εξετάσουν αυτά, δηλαδή η δική μας νομοδότηση. Κατανοώ, Πρόεδρε, ότι πρέπει να υπάρχουν προδιαγραφές εργασίας, ε, προϋποθέσεις, συνθήκες εργασίας και αυτά ισχύουν και για τις μεταφορές και πρέπει να μπουν στη δική μας γνωμοζότηση. Κοινωνικό ντάμπινγκ, η οδηγή φορτηγών, όλα αυτά είναι μεγάλο θέμα. Και ε, δεύτερο, θα πρέπει να μπει κάτι για το ESDS, το Σύστημα Διευθέτησης και Επίλυσης Διαφορών Επενδυτή Κράτους. Ε, αυτό αφορά και τις δημόσιες προμήθειες στις ΗΠΑ Πολιτείες και είναι άρρηκτα συνδεδεμένο με τη Συμφωνία TTIP. Αυτά εισαγωγικά για το θέμα. Ελπίζω να ακούσω σχόλια από τους συναδέλφους για να τα επεξεργαστούμε και πάλι με τη γραμματεία την οποία και πάλι ευχαριστώ για την υποστήριξη. Θα εμβαθύνουμε λοιπόν και η ψηφοφορία είναι την άλλη 5η το πρωί 26 του μηνός Μαρτίου. Σας ευχαριστώ πολύ. Danke sehr. Jetzt. Ευχαριστώ πολύ. Ο Ισμαήλ Ερτούκ προσωπεί τον κύριο Λάιχφριτ. Ja, Schönen guten Morgen. Καλημέρα σας λέει ο κύριος Ερτούκ. Ich habe nämlich äh, in die falsche Richtung geguckt, lieber Wim. Αγαπητέ Wim, κοίταγα σε λάθος κατεύθυνση, <laughs> οπότε γυρνάω σε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, ε, ευχαριστώ. Ε, ο κύριος Λάιχτφριτ κολλείεται και τον αντικαθιστώ εγώ σήμερα. Θα σας παρουσιάσω τη θέση της ομάδας των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών. Μπορώ να σας πω ότι από πλευράς μας εμείς σε ό,τι αφορά τη συμφωνία TTIP με τις Ηνωμένε Πολιτείες, τη θεωρούμε ε, σημαντική ευκαιρία. Αλλά θα πρέπει να τονίσουμε την ευκαιρία αυτών ε, τη σημασία των μεταφορών ε, και να τονιστούν ιδιαίτερα ορισμένα θέματα. Καταρχήν συμφωνούμε και είμαστε ικανοποιημένοι με την γνωμοδότηση και θέλουμε να ευχαριστήσουμε και εγώ προσωπικά τον εισηγητή μας τον κύριο Κάμπ για την εργασία του και επίση ε, αυτό όμως δεν αλλάζει τίποτα στο γεγονός ότι θα πρέπει να εκπονήσουμε συμβαστικές τροπολογίες. Ε, βασικοί ε, κανόνες και προδιαγραφές του Διεθνούς Γραφείου Οργανισμού Εργασίας είναι κάτι σημαντικό. Προδιαγραφές εργασίας και πρότυπα και η εφαρμογή τους δεν αναφέρονται καν στις συμβαστικές προτάσεις, ούτε για τις κυρώσεις κάνει λόγο εισηγητή σε περίπτωση παραβίασης, ούτε για το κανονιστικό πλαίσιο δεν αναφέρεται ρητά η απαγόρευση της μείωσης ή των εκπτώσεων σε ό,τι αφορά τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές. Και για το ISDS, το σύστημα επίλυσης διαφορών επενδυτή κράτους, μπορεί να έχει σημασία και για τις μεταφορές είναι πολύ σαφή η θέση των σοσιαλδημοκρατών. Θεωρούμε ότι σε μια συμφωνία Ευρώπης Ηνωμένων Πολιτειών δεν έχει ε, καμία θέση μια τέτοια ρήτρα. Για τις υπηρεσίες θα θέλαμε πιο ισχυρή διατύπωση, ιδιαίτερα ε, να μην υπάρχουν αρνητικοί κατάλογοι, ε, υβριδικές ε, ρήτρες και ε, θα πρέπει να υπάρχουν ε, ε, Ε, επίσης ευκαιρίες και δυνατότητες να ανοίξουν ε, κάποιες αγορές παροχής υπηρεσιών και άλλες και να μην επηρεάζονται σε καμία περίπτωση από εμπορικές συμφωνίες. Ε, έχουμε προτάσεις, θα τις δώσουμε στον εισηγητή, ελπίζουμε να μπουν στο συμβιβασμό και αν συμβεί κάτι τέτοιο προσβλέπουμε σε μια καλή γνωμοδότηση στον εισηγητή που είναι αρμόδια επιτροπή τη ουσία όπως γνωρίζετε Επιτροπή Διεθνούς Εμπόριου. Αυτά από τους σοσιαλιστές. Ευχαριστώ πολύ, ευχαριστώ και εγώ η Τζάκη Φώστερ. Ε, Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Θέλω να ευχαριστήσω τον εισηγητή μας, ε, τον κύριο Φάντεν Κάμπ. Νομίζω ότι είχαμε μια επικοδομητική συνάντηση και κάποια από τα σημεία τα οποία συζητήθηκαν εκεί νομίζω ότι λαμβάνονται υπόψη στις ε, αρχικές συμβαστικές προτάσεις και το θέμα βέβαια ήταν μετά για τον εισηγητή να προσπαθήσει κάπως να τα συμβιβάσει όλα αυτά και να τα διατυπώσουμε με τον σωστό τρόπο. Εμείς θεωρήσαμε ότι δίνεται στο 1α πολύ έμφαση σε ορισμένες κοινωνικές πτυχές. Φυσικά και στηρίζουμε βέβαια ε, τις καλές συνθήκες και όρους εργασίας, αλλά εδώ ε, είμαστε Επιτροπή Μεταφορών. Η Επιτροπή Απασχόληση σίγουρα έχει τα δικά τη θέματα και θα κάνει τις δικέ προτάσει. Αυτό είναι το πρώτο σημείο. Αλλά στο 1α είναι Θετικέ τέλο πάντων οι αλλαγές τις δεχόμαστε. Σε ό,τι αφορά το 3, το έχουμε συζητήσει. Αν δει κανεί τα θέματα ιδιοκτησία, ε, σε ό,τι αφορά τις σχέσεις Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, και η ε, ακόμα έχουν γίνει κάποιες βελτιώσεις, αλλά πολλά απομένουν να γίνουν. Στο καμποτάζ ή τις ελευθερίες τώρα, Έχουμε κάποια απόψεις και το είπαμε και στη συνάντηση με τους Κιώδης. Είναι αμφίδρομο. Οι αμερικανικές αεροπορικές εταιρείες δεν παίρνουν τις ελευθερίες που λέμε εμείς ότι δεν μπορούμε να έχουμε στις ΗΠΑ. Γι' αυτό γίνονται και συμμαχίες άλλωστε. Γίνεται μεν αναφορά στο ότι δεν μπορούν κάποιες εταιρείε ε, να κάνουν κάποια πράγματα στη ΣΥΠΑ, αλλά ούτε στην Ευρώπη δεν μπορούν να τα κάνουν. Άρα πρέπει να αναφέρουμε τα πραγματικά περιστατικά. Πιο πολύ είναι το θέμα του ελέγχου. Ουσιαστικά μιλάω για τις ε, υπηρεσίες αεροπορικών, για τις συμφωνίες αεροπορικών υπηρεσιών. Πάντως, έχει κάνει μια γνήσια προσπάθεια ο ε, για να συμβιβάσει η αρχική του έκθεση ήταν πολύ καλή, έχει εστιάσει στις σωστές ε, πτυχές, σωστούς τομείς κατ' εμάς. Αυτά από πλευρά CCR. Και ευχαριστώ και πάλι τον εισηγητή. Γκεζίνε είναι τώρα, λέει ο πρόεδρος. Ευχαριστώ πρόεδρε, ευχαριστώ και εγώ τον Βιμ Καμπ. Τον γνωρίζει, έχω πει από την αρχή ότι είναι πάρα πολύ καλή, θαυμάσια, υπέροχη η γνωμοδότησή του. Γι' αυτό δεν έχω κάνει ούτε μία τροπολογία παρακαλώ. Διότι συμφωνούσα 100% με το συντάκτη της γνωμοδότησης. Τώρα έχουν υποβληθεί κάποιες τροπολογίες και από τη δική μου πολιτική ομάδα, Ντομινίκ Ρικέ ας πούμε, έχει κάνει μερικές. Ε, υπήρχαν ήδη συμβιβασμοί, του οποίου διαπραγματευτήκαμε και ήταν πάρα πολύ καλή και η προεργασία που είχε κάνει, Βιμ. Πρέπει να το πούμε και αυτό. Έχει συμπεριλάβει προτάσει διαφόρων πολιτικών ομάδων. Προσωπικά πιστεύω ότι το κείμενο είναι πάρα πολύ ισόρροπο. Δεν θα ήθελα να αλλάξουμε κάτι ε, αυτή τη στιγμή. Στην αρχή προτάθηκε κάτι για τεχνολογία, δεν διαφωνεί κανείς το 1α. Επίσης ε, γίνεται λόγος για την προστασία των προσωπικών δεδομένων και της ιδιωτικής ζωής. PNR ήταν κάτι που συζητήθηκε, αν θα ε, πρέπει να το πούμε. Καλό είναι αυτό που λέμε, αλλά από εκεί και πέρα Κύριε Ερτούκ, δεν πιστεύω ότι θα πρέπει να μιλήσουμε για το ILO. Είμαι πολύ υπέρ των δικαιωμάτων των εργαζομένων και στη χώρα μου είχα εργαστεί για αυτά τα θέματα. Αλλά επειδή γνωμοδοτεί κάθε επιτροπή, ας αρκεστούμε εμείς και ας περιοριστούμε στα δικά μας χωράφια των μεταφορών. Το έχουμε ξαναπεί αυτό για τη σημασία των εργαζομένων, για τα συνδικάτα, για τις διαπραγματεύσεις, όλα αυτά τα αναφέρουμε. Τι δουλειά έχει ο ILO. Θέλουμε να έχουμε καλές συνθήκες εργασίας μέχρι εκεί. Τώρα, στο 2 ε, για να συμπεριληφθεί το σύστημα διευθέτησης διαφορών επενδυτή κράτους, ISDS, ε, έχει συμπεριληφθεί με τρόπο ισόρροπο και μια σωστή ε, διατύπωση. Το έχουμε συζητήσει, αφορά και τις μεταφορές, βεβαίως θα πρέπει να αναφέρεται, αλλά με αυτόν τον τρόπο. Παρόλο που είχαμε συμφωνήσει ότι για το τι γενικά θα μπορούσε να πει κανείς πολλά πράγματα γενικά, αλλά δεν μας ενδιαφέρουν τα γενικά, μας ενδιαφέρουν τα ειδικά. Γνωμοδοτούμε ως Επιτροπή Μεταφορών. Αυτό με τις αεροπορικές εταιρείες μου αρέσει, γιατί ε, είμαστε πάντα ρηγμένοι στις συμφωνίες εμείς οι Ευρωπαίοι για τα αεροπορικά. Δεν είμαι τόσο αφίλη που να πιστεύω ότι θα κάνουμε τώρα το μεγάλο άλμα ή το μεγάλο βήμα, αλλά ας το δοκιμάσουμε, ας το προσπαθήσουμε για να διαπραγματευόμαστε επί ώρες, γιατί συνήθω μας ρίχνουν Ηνωμένες Πολιτείες. Το 5 έχουμε βάλει κάτι που ζήτησε ο Ντομινίκ Ρικέ, πόσο δύσκολο είναι για μας να διαπραγματευόμαστε, το έχουμε πει, γιατί εμείς έχουμε ε, ε, ένα σύστημα, ας πούμε, ομοσπονδιακό, είμαστε πολλές χώρες, οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι μία χώρα. Ε, πάντως, στη συνεδρίαση των σκιωδών εισηγητών. Βιμ, πραγματικά ήταν πολύ καλό το κλίμα και το αποτέλεσμα και το προϊόν μου αρέσει πάρα πολύ. Kiitoksia puheenjohtaja. τα μάμπου. Μαρία Κίλε. Ναι. Ευχαριστώ πολύ. Την Άνια Γκονθάλες Μπενάλβες εκπροσωπώ. Θα τα πω αγγλικά όμως γιατί μου τις έδωσε στα αγγλικά αυτές τις ε, σημειώσεις. που δεν μπορούσε να είναι παρούσα. Θέλει να ευχαριστήσει τον κύριο Κάπ για το επικοδομητικό του έργο. Διαβάζω τώρα τι έγραψε. Όπω έγινε το 1988, όταν τον κοινό και σταμάτησε η διαπραγματεύση για την πολυμερή συμφωνία, ε, θα πρέπει τώρα να κάνουμε προσπάθειες για να αποκαλύψουμε και να παρουσιάσουμε ε, την πραγματικό πρόσωπο αυτής της ε, συμφωνίας, της Ιρλανδικής Συμφωνίας της και του Εμπόριο, TTIP. Η κρίση η οποία πλήττει ολόκληρη την Ευρώπη φαίνεται να είναι πρόσφορο έδαφος, ε, ένα πρόσχημα ότι δηλαδή τάχα θα υπάρξει ανάκαμψη οικονομίας και δημιουργία απασχόληση με αυτή τη συμφωνία. Αν δηλαδή εφαρμοστεί ένα νέο ρυθμιστικό πλαίσιο που είναι κομμένο και ραμμένο στα μέτρα των πολυεθνικών. Προωθείται ένα οικονομικό μοντέλο όπου η οικονομική ολιγαρχία αποκτά και εκμεταλλεύεται την πολιτική εξουσία για να εκμεταλλευτεί τους πόρους και τον πλούτο που ανήκουν όμως όλους τους πολίτες. Αυτή η συνθήκη όμως δεν φετερίζεται μόνο πολιτική εξουσία, αλλά και προωθεί ένα μηχανισμό για την επίλυση διαφορών μεταξύ κυρίαρχων κρατών και επενδυτών. Αυτό το λεγόμενο ISDS, που είναι αντιδημοκρατικό, αντιδημοκρατικός μηχανισμός και δεν μπορούμε να τον αποδεχθούμε και στον τομέα των μεταφορών, όπως και σε άλλους τομείς της οικονομίας, κανονισμοί οι οποίοι είναι υπέρ των μεγάλων εταιριών, ουσιαστικά δημιουργούν αολιγοπόλια και οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις ε, λόγω αυτού ε, καταφεύγουν σε μια επισφαλή τακτική αυτή της εξωτερικής ανάθεσης. Επίσης υποβαθμίζονται τα πρότυπα και οι δημόσιες υπηρεσίες που είναι πολύ σημαντικές όμως στον τομέα των μεταφορών για την κοινωνική και την εδαφική συνοχή. Δεν μπορούμε να δεχθούμε συμφωνίες ελεύθερων συναλλαγών που θα οδηγούν σε αύξηση των ανισοτήτων και των επισφαλών θέσεων εργασίας, με ανασφάλεια ή υποβάθμιση του περιβάλλοντος. Όσο διαπραγματεύονται ε, εγκρυφό και παραβίστο οι διάφοροι αυτή τη συμφωνία, δεν θα μπορέσει να καταλάβει ο κόσμος περί τίνος πρόκειται. Αλλά πριν ληφθεί οποιαδήποτε απόφαση θα πρέπει να έχει ενημερωθεί και η κοινή γνώμη. Δεν θα πρέπει να βαθμιστεί το περιβάλλον, ούτε να περιοριστούν οι ελευθερίε και τα δικαιώματα των πολιτών. Μια τέτοια συμφωνία δεν πρόκειται να την εγκρίνω. Αυτά είπε η Τάνια. Ευχαριστώ. Η Καριμά Ντελή, που μόλι κατέφθασε, έχει το λόγο εξ ονόματο τη ομάδα τη. Ευχαριστώ, Πρόεδρε εξ ονόματος της ομάδας μου να ζητήσω συγγνώμη εκ μέρους του κυρίου Μπάς Εκχαλτ, ο οποίος δεν μπορεί να είναι μαζί μας. Η πολιτική γραμμή αυτού του σχεδίου γνωμοδότησης συμπεριλαμβάνει πολλές συμβαστικές λύσεις που είναι μάλλον θετικές, ιδίως για την ομάδα μας. Είτε πρόκειται για τις περιβαλλοντικές πτυχές, είτε για τα πρότυπα των οχημάτων, των αυτοκινήτων, αλλά και όλα τα πρότυπα για την αμοιβαιότητα των δικαιωμάτων, για την εσωτερική αγορά, τα δικαιώματα των επιβατών, την ε, χορύπανση ή ό,τι αφορά τα αεροδρόμια. Επίσης, μπορούμε να πούμε ότι κάποια σημεία θα πρέπει να ενισχυθούν όταν γίνεται λόγος ε, ιδίω για την διαφάνεια ή όταν μιλάμε για τα δικαιώματα των πολιτών. Εκεί πρέπει να τονίσουμε, την, ε, να ενισχύσουμε τη σημασία στη διατλαντική συνθήκη της ε, διάστασης των μεταφορών. Πρέπει να ενισχυθούν τα σημεία που αφορούν την ασφάλεια, το κλίμα και το περιβάλλον. Και πρέπει να, αποδει... να δείξουμε ότι η οικονομική ανάπτυξη χρειάζεται βέβαια, αλλά με θέσει απασχόληση βιώσιμε. Όταν μιλάμε για βιωσιμότητα των θέσεων απασχόληση, εννοούμε για ε, μιλάμε για ποιότητα, για αξιοπρέπεια. Και επίση πρέπει να δοθεί έμφαση σε αυτό που εμεί αποκαλούμε το σύνολο των προτύπων για την ε, διάσταση των αυτοκινήτων, των οχημάτων. Όταν ε, μιλούμε για εκπομπές διοξιδίου του άνθρακα δεν πρέπει να λησμονούμε ότι αυτό σχετίζεται με την διάσταση των μεταφορών. Ευχαριστώ πρόεδρε. Ευχαριστώ πολύ. Η Ρόζα Νταμάτο. Ε, Ευχαριστώ πρόεδρε. Ευχαριστώ την εισηγήτρια για τις, τον ε, συγκεκριτή για τις τροπολογίες που υπέβαλε. Αλλά πρέπει να πω ότι έχουμε μια διαφωνία επί της ουσίας με την ε, συμφωνία TTIP, ιδίω για τη διάσταση των μεταφορών. Είναι πολύ σημαντικό και ιδίω ό,τι αφορά τον μηχανισμό επίλυση διαφορών μεταξύ κρατών και επενδυτή. Ε, οι τροπολογίε εκφράζουν ε, κάποιε βελτιώσει, αλλά πολύ ήπιε. γι' αυτό θέλουμε να υπάρξει πλήρη αποκλεισμό των ρητρών ευθύε. Γιατί, Γιατί ο μηχανισμός αυτός ε, ουσιαστικά επιβάλλει διακριτική μεταχείριση ευνοεί του ξένου επενδυτέ ει βάρο των εσωτερικών, των εθνικών. Δίνει έμφαση στα δικά του ειδικά προνόμια που άλλα μέρη της κοινωνίας δεν τα διαθέτουν και δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη. Η διακριτική μεταχείριση υπέρ των ξένων επενδυτών μπορεί να καταστρέψει την ισότητα στον ανταγωνισμό που για την ώρα υπάρχει μεταξύ εθνικών και αλλαδαπών επενδυτών. Δεν θα υπάρχει καμία βεβαιότητα δικαίου και με επιχειρηματολογία για θέματα όπω οι βοήθειε ή οι δημόσιοι διαγωνισμοί. Άρα, Υπάρχει και ένα θέμα διαφάνεια ό,τι αφορά αυτό το μηχανισμό. Οι διαιτητέ θα αποφασίζουν κατά πόσον υπάρχει ανάγκη να ε, προστατεύονται πληροφορίε προστατευμένε ή χαρακτηρισμένε ή απόρριτε. Εκεί θα πρέπει να ε, φροντίσουμε οι συνθήκε να ισχύουν και να επιβληθεί η προσφυγή στα παραδοσιακά δικαστικά συστήματα. Και βάσει των προτάσεων τη Επιτροπή δίνω παραδείγματα τώρα. Ε, Φαντάζομαι ότι το γνωρίζετε, οι περιπτώσεις ε, της υπόθεση Φίλιπ Μόρι και η απόπειρες τη να προβλέψει νομοθεσία κατά των προϊόντων καπνού ή η ε, το, πρωινό, το προσωρινό μνημόνιο κατανόηση για την υδρορογμάτωση στο Κεμπέκ, όλα αυτά δείχνουν ότι ε, υπήρξαν κάποιε αποφάσει για απολύσει χωρί να δοθεί ε, βάση στην ουσία του κειμένου τη Επιτροπή. Η πρόταση τη Επιτροπή λέει ότι οι διαιτητέ αποφασίζουν. Ο μηχανισμό ουσιαστικά πλήττει το δικαίωμα των κρατών να προβλέπουν κανόνε. Και αυτό θεωρούμε ότι πραγματικά ε, υπονομεύει τις κυβερνήσεις. Με κυρώσεις που μπορεί βάσει των νέων νόμων να υπονομεύουν και να βλάπτουν το δημόσιο δίκαιο. Οι, τα αποτελέσματα των διαβουλεύσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής δεν επιτρέπουν ε, να καλύπτεται η απασχόληση και δεν υπάρχει και κανένα, ε, καμία σοβαρή μελέτη αντικτύπου για την επίδραση του μηχανισμού αυτού, του ISDS, στις μεταφορές. Οπότε, πρέπει να αποκλειστεί μέχρι να υπάρξει μια διεξοδική και αξιόπιστη μελέτη για τον μηχανισμό αυτό και να, τον έχουμε συζητήσει, να την έχουμε συζητήσει μάλλον και στο Κοινοβούλιο. Ευχαριστώ. Κυρία Ευχαριστώ πολύ. Θέλω να ευχαριστήσω τον εισηγητή. που έχει συμπεριλάβει συγκεκριμένε επιτυχίες για τις μεταφορές που δεν νομίζω ότι είναι και πτυχές άσχετες με τη διαπραγματευσή της όλης αυτής συμφωνίας. Εργασιακές συνθήκες, ε, περιβάλλον... Εγώ δεν νομίζω ότι θα έπρεπε να είναι σε κάποιο άλλο σημείο, το έχουμε πει πολλές φορές. Ένα από τα γενικά προβλήματα του τομέα των μεταφορών, όχι μόνο σε ευρωπαϊκό αλλά και σε παγκόσμιο επίπεδο, είναι ακριβώς οι εργασιακές συνθήκες το ότι δεν είναι ελκυστικές οι συνθήκες εργασίας στον τομέα των μεταφορών. Και αυτό δημιουργεί κινδύνους, απειλές για την ασφάλεια, τα δικαιώματα των επιβατών, την ασφάλεια, ακόμη και για την ανάπτυξη. Άρα το να μιλάμε για τον περιβαλλοντικό αντίκτυπο νομίζω είναι ε, σωστό. Έχω καταθέσει τροπολογίες με τις οποίες ζητώ σε καμία περίπτωση να μην δεχθούμε η συμφωνία να μειώσει τα περιβαλλοντικά και κοινωνικά πρότυπα που ισχύουν στην Ευρώπη. Άλλωστε αυτό περιμένουν και οι εργαζόμενοι στον τομέα των μεταφορών. Το ίδιο ισχύει με το δικαίωμα των επιβατών. Δηλαδή στην Ευρώπη επιτέλους σιγά σιγά καταφέραμε να εδρεώσουμε μια νομοθεσία και αυτό ήταν και αποτέλεσμα πολύ καλής ε, διαπραγμάτευσης με τους διάφορους κλάδους και όλους τους εμπλεκόμενους ε, φορείς για τα δικαιώματα των επιβατών. Είναι λοιπόν πάρα πολύ σημαντικό τώρα να διατηρηθούν σε επίπεδο αυτό και τα δικαιώματα αυτά. Και αντίστροφα, στην, ε, στο πλαίσιο της αντιπροσωπείας μας ε, με την Άσκτον με την Αμερική που είχαμε στην Ουάσιγκτον, εκεί μιλήσαν και για τα, για το, τα πληρώματα ε, θαλάμου επιβατών. Δεν μπορούμε να δεχθούμε να υπάρχει κοινωνικό dumping και αυτό να χρησιμοποιείται ως στοιχείο του ανταγωνισμού και εργασιακές συνθήκες το ίδιο για το μισό αυτό αυτός της αεροπορίας. επίση έχω άλλε δύο τροπολογίε Είμαι αφορά την ασφάλεια των μεταφορών. Υπάρχουν εξελίξεις και ανάπτυξη και από τις δύο πλευρές. Προστασία δεδομένων, θα το δούμε και αυτό βέβαια. Να δούμε τι μπορεί να γίνει. Να είναι σαφέ βέβαια το τι γίνεται με την προστασία των ε, δεδομένων, πάντα σύμφωνα με τα ευρωπαϊκά πρότυπα και δημόσιες υπηρεσίες. Δεύτερο. Εδώ δεν είναι απαραίτητο μόνο να προστατεύσουμε τις μας υπηρεσίες, αλλά να μην απειληθούν ή να υποβαθμιστούν αυτές οι υπηρεσίες σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Λόγω μια τελείως διαφορετική αντίληψη που επικρατεί για δημόσιες υπηρεσίες της είπα. Yes, I wouldn't normally uh, come in after a colleague. Δεν ήθελα να πάρω το λόγο μετά τη συνάδελφο, αλλά η κυρία Γιάλα Σέντερ έλεγε για υποβολή τροπολογιών. Οι συμβαστικέ τροπολογίε που συζητήσαμε με τον εισηγητή κάτι δεν έχουν ε, καλύψει νομίζω. Δεν είμαι βεβαία λοιπόν. Έχουμε 78 τροπολογίε περίπου και έχουμε καταλήξει σε συμβαστικέ λύσει. Τώρα τι θέλετε να, βάλουμε κι άλλες να υποβάλουμε και άλλε τροπολογίε ή κάτι δεν κατάλαβα. Νόμιζα ότι μιλούσατε για επιπλέον τροπολογίες. Κάτι ίσως να μην κατάλαβα από τη μετάφραση. Σας ευχαριστώ για τη διευκρίνηση. Ακούστε. Ναι, ε, δεν τις έχετε διαβάσει μάλλον ε, και γι' αυτό τις είπα εγώ. Και αυτό με ανησυχεί. Δηλαδή κάνω τις συμβαστικές ε, τροπολογίες χωρίς να έχετε διαβάσει τις ε, δικές μου παραδείγματος χάρη τροπολογίες. Εντάκη Φώστερ, άμα είσαι καινούριο μέλος στο κοινοβούλιο, δεν έχει μάθει ακόμα τους κανόνες. Η Κριστίν Γοβεντολόν έχει το λόγο, παρακαλώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε, και ευχαριστώ τον συγητή για τη δουλειά του, που πραγματικά συζήτησε και ήρθε σε διάλογο με όλες τις ομάδες. Ήταν πολύ σημαντικό αυτό. Το έχω ξαναπεί όταν πρώτο συζητήσαμε τη συμφωνία TTIP ότι είναι σημαντικό η Ευρωπαϊκή η Επιτροπή Συγγνώμη Μεταφορών να ασχοληθεί με το συμφωνία αυτή, ιδίω για τη διάσταση των μεταφορών. Πολλά επιχειρήματα ακούσαμε και από του συναδέλφου, ε, κυρίως από την κυρία Γιάλα Σέντερ, και είναι σαφέ ότι δεν θέλουμε η συμφωνία TTIP να αντίκειται στο γενικό συμφέρον και να, δίνει, ε, να ευνοεί ουσιαστικά τους, ε, τις ευρωπαϊκές εταιρείες και τους υπαλλήλους τους. Για την δική μας την ομάδα δεν υπάρχει κανένας λόγος στη συμφωνία να συμπεριλαμβάνεται η ιδιωτική διατησία, διότι ε, η εθνική δικαιοδοσία και οι δημοκρατικές αρχές επί των οποίων βασίζονται οι κοινωνίες μας. Η τροπολογία 18 που συλλαμβάνεται στην ε, έκθεση και καλεί την Επιτροπή να, να σεβαστεί τα αποτελέσματα των δημόσιων διαβουλεύσεων για το μηχανισμό ISDS είναι σημείο κλειδί τη έκθεση. Επίσης, πρέπει να βεβαιωθούμε ότι η συμφωνία TTIP δεν επιβάλλει ε, δεσμευτικούς κανόνες τα κάτι μελη και τις περιφερειακές αρχές να απελευθερώσουν ή ιδιωτικοποιήσουν τις δημόσιες υπηρεσίες, κάτι που θα ήταν καθοριστικό για την προσφορά υπηρεσιών μεταφοράς ε, ποιότητας και που να είναι προσβάσιμη σε όλους. Κατά τρίτον, βάσει τη αρχή τη αμοιβαιότητα, πρέπει να καλέσουμε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να δώσει ιδιαίτερη προσοχή στου περιορισμού και τι διακριτικέ μεταχειρήσει που ισχύουν στι ΗΠΑ ω προ την πρόσβαση στην αγορά των επενδυτών. Η πρόσβαση στι δημόσιε προμήθειε και η πρόσβαση των αεροπορικών εταιριών είναι ευαίσθητα ζητήματα, επί των οποίων πρέπει να υπάρξει μια σαφή δέσμευση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Για να ολοκληρώσω και πιο συνολικά, ιδίω για να έχουμε καλή τήρηση των δεσμεύσεων που έχουν ζητήσει οι Ευρωβουλευτέ, είναι πρωταρχή σημασία διαδικασία να υπάρξει μεγαλύτερη διαφάνεια από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τι ανεξελίξει διαπραγματεύσει. Ευχαριστώ. Κύριε Σκόχ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Όπως και όλοι σας, και εγώ κατακλείζομαι από τα ίδια mail και υπογραφές που με καλούν να ε, καταψηφίσω συλλήβδιν και να απορρίψω το TTIP. Φυσικά δεν θα το πράξω. Ευχαριστώ το συντάκτη νομοδότησης για την πολύ καλή του πρόταση έχουν πολύ μικρές συμπληρώσεις. Η διαπραγματευτική εντολή δεν θα πρέπει να περιορίζεται μόνο στις μεταφορές αλλά και στον τουρισμό και την εφοδιαστική logistics και να έχουμε μια κριτική ματιά. Επίσης, ε, πολλοί ομιλητέ αναφέρθηκαν στις δικές μας αεροπορικές εταιρείες που είναι σε μειονεκτική θέση. Δεν θέλω να επανέλθω παρόλο που έχω κάνει σχετική τροπολογία και τρίτον ο προστατευτισμός. Ε, αγαπητέ Βιμ, ε, ότι θα πρέπει να τον αναφέρουμε. Εγώ δεν θέλω μόνο να τον αναφέρουμε, αλλά και να τον καταργήσουμε, δηλαδή λίγο πιο οξία η διατύπωση. Η Μαρή Κριστίνα Ανότ. Κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, όπως και στην προηγούμενη συνεδρίαση της Επιτροπής μας, επαναλαμβάνω τη διαφωνία του Front National σε οποιαδήποτε συμπερίληψη νέων θεμάτων, ιδίω ό,τι αφορά τι μεταφορέ, τι διαπραγματεύσει ε, μεταξύ Ευρωπαϊκή Ένωση και ΗΠΑ για την εταιρική σχέση, τη διατλαντική. Ε, Προφανώ ε, δεν συμφωνούμε με τι τροπολογίε που θέλουν να διευρύνουν ακόμη την πρόταση για το μηχανισμό επίλυση και ιδίω για τα θέματα τουρισμού. Θα στηρίξουμε τι τροπολογίε 8 και 76 των συναδέλφων Νταμάτο και Αγιούτο. Από μήνε το Front Φινάλ καταγγέλει τι απειλέ που η συμφωνία TTIP μπορεί να ε, ε, σημαίνει για τα εθνικά συμφέροντα, την εθνική κυριαρχία και του λαού, ιδίω για να προσπιστούν τα συμφέροντα των πολυεθνικών. Είναι πραγματικά θλιβερός ο προστατευτισμός των Ηνωμένων Πολιτειών και επιτέλους θα πρέπει να σταματήσουν οι στρεβλώσεις ανταγωνισμού που ε, έχουν δεσμενείς επιπτώσεις για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν νομίζω ότι μπορούμε να υποχωρήσουμε ε, απέναντι στους ε, Αμερικανούς και ότι, θα πρέπει, και ότι κάτι τέτοιο θα πρέπει να το επιτρέψουμε. Θα πρέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη-μέλη να πραγματιστούν από τις Ηνωμένες Πολιτείες και να εξοπλιστούν με τα απαραίτητα εργαλεία ιδίω ό,τι αφορά την ε, τελωνιακή, τα τελωνιακά για να προστατεύουν και τη δική του οικονομία. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Να ευχαριστήσω τον ε, εισηγητή. Οι μεταφορέ είναι βεβαίω μια πολύ σημαντική διάσταση όλη αυτή τη συμφωνία και το κοινωνικό ντάμπινγκ είναι μέγιστη απειλή για την ε, ασφαλεία μα. Βλέπετε τα αποτελέσματα στις μεταφορές γενικότερα στην Ευρώπη αυτή τη στιγμή. Αλλά για το καμποτάζ ας πούμε πρέπει να υπάρξουν αλλαγές. Και εγώ θέλω να είμαι σαφής και ειλικρινής. Είναι τελείως ανοησίες αυτά που συμβαίνουν. Ε, απάτες, κατάχρηση, καταχρηστική ερμηνεία της Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας. Εάν μιλήσουμε για προσετακτισμό, να σας πω κάτι που άκουσα πρόσφατα είναι προστατευτισμός να ισχύουν αξιοπρεπή πρότυπα και κανόνες. Όχι. Προφανώς και όχι. Δεν θα έπρεπε να επιτρέπουμε την εκμετάλλευση των ανθρώπων στον τομέα των μεταφορών. Το ίδιο και για τις αεροπορικές ε, μεταφορές. Όλο και περισσότερα γραφεία απασχόλησης ε, είναι αυτά που, ε, στα οποία τρέχουν οι εταιρείε για να παρακάμψουν την νομοθεσία την εργασιακή. Αυτό θα πρέπει λοιπόν να ισχύει για τα πληρώματα ε, της καμπίνας επιβατών και ένα σωρό άλλα ζητήματα ανακύπτουν εδώ. Θα πρέπει να υπάρχουν αυστηρότερες ε, προδιαγραφές σε πολλά επίπεδα. Όμως η συζήτηση πρέπει να παραμείνει ανοιχτή για να μπορέσουμε να βελτιώσουμε τη συμφωνία. Πάντω ο εισηγητή έχει κάνει εξαιρετική δουλειά. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Είναι βέβαια για μας πολύ κομβικό αυτό το θέμα και η Συμφωνία Ελευθέρων Συναλλαγών με τις Ηνωμένε Πολιτείε μας απασχολεί πολύ. Έχει σημασία η Επιτροπή Μεταφορών να γνωμοδοτήσει, αλλά το είπε και ο εισηγητής, Βιμ Βαντεκάμπ και το ξεκαθάρισε, θα πρέπει να επικεντρωθεί στα δικά της θέματα η Επιτροπή μας, σε θέματα μεταφορών και σε θέματα τουρισμού. Αυτά να είναι στο προσκήνιο. Και είναι σημαντικό βεβαίως να αποφανθούμε και να επικεντρωθούμε σε αυτά τα θέματα και να δούμε τι γίνεται με το σύστημα εμπορίας εκπομπών ρήπων, τι ε, γίνεται ε, με τις θαλάσσιες μεταφορές, ε, έχουν αντίστοιχε καταστάσεις να αντιμετωπίσουν και οι Αμερικανοί για τους ελέγχου, Τι γίνεται με τον έλεγχο του κράτους λιμένα, ε, τι γίνεται με τη διεκπαιρέωση, πώς γίνονται οι υπηρεσίε στα λιμάνια και τα αμερικανικά και τα δικά μα, Γιατί αυτά θα πρέπει να μας απασχολήσουν αυτή τη συμφωνία, θαλάσσιε μεταφορές. Δεν έχουμε εκεί αυτοκίνητο δρόμους, έχουμε τον Ατλαντικό. Ε, καταλαβαίνετε ότι είναι σημαντικό αυτό το θέμα και μας απασχολεί πάρα πολύ και εγώ θέλω να από ότι είμαστε υπέρ όλων των δικαιωμάτων και των εργαζομένων και ό,τι άλλο θέλετε, αλλά να το αφήσουμε αυτό στα χέρια των αρμοδιών επιτροπών. Υπάρχει μια επιτροπή που λέγεται απασχόληση και κοινωνικών υποθέσεων και θα γνωμοδοτήσει και αυτή. Λοιπόν, θα κάνουμε καλά να ακολουθήσουμε τη συμβολή του Βανταγκάμπ, να υποστηρίξουμε την καλή του γνωμοδότηση και να εστιάσουμε στα δικά μας θέματα που είναι και σημαντικά, επαναλαμβάνω. Ο Πρόεδρος θέλω να θυμίσω ότι όταν πήγαμε στις Ηνωμένες Πολιτείες, στο τέλος ε, με το ταξί πέρασα από ένα διοικητικό κτίριο που ήταν το εμπορικό επιμελητήριο, δεν ξέρω, είχε μια μεγάλη πινακίδα και έγραφε «Fair conditions with our partners». Ε, να έχουμε δίκαιες ε, συνθήκες με τους εταίρους μας. Ναι, αλλά δεν το έχουμε στις αερομεταφορές ή κάπου αλλού. Το τονίσαμε εμείς, δεν υπήρχε καμία προθυμία να τα αλλάξουν. Μας είπαν ότι υπάρχουν ε, συμφωνίες, γιατί να τις αλλάξουμε εις βάρος μας. Το κατανοούμε, αλλά ε, αν είναι προς δικό μας μειονέκτημα, για να μην προσπαθούμε εμείς να το αλλάξουμε. Ενδιαφέρον αυτό. Σήμερα στην εφημερίδα Τάκε Σπίγκελ του Βερολίνου είχε ένα άρθρο για το TTIP και λέει για την ε, διαδικασία αυτή την εξοδικαστική στην ε, Αυστρία, έχουν ε, τώρα προσφύγει στα δικαστήρια ε, γιατί ε, η Φίλιπ Μόρις έχει προσφύγει κατά της κυβέρνησης της Αυστραλίας λόγω των προεδοποιήσεων που έχουν βάλει στα πακέτα των τσιγάρων και έχει χάσει λεφτά η Φίλιπ Μόρις και τα ζητάει από την κυβέρνηση της Αυστραλίας και τα έχουν υπολογίσει κιόλα. Σα δίνω παραδείγματα. Δεν μου επιτρέπετε να πω παράδειγμα. Για ποιο λόγο. Ε, εγώ έχω εγγραφεί στην ημερήσια διάταξη ως ομιλητή. Δεν έχει καμιά σχέση, λέει κάποιο. Φυσικά και έχει σχέση. Αυτό είναι το αποφασιστικό θέμα. Άλλη είναι η συζήτηση για ε, τις συμφωνίες εμπορικών ε, συναλλαγών αν δεν υπάρχουν ε, εξάρτητοι διαιτητές. Διότι είμαστε δύο κράτη ή ξέρω εγώ κρατικές οντότητες που έχουμε ανεξάρτητη δικαιοσύνη. Δεν χρειάζεται έξτρα διαιτησία. Θα πρέπει να βρούμε ένα συμβιβασμό και δεν μου επιτρέπετε να το πω επειδή είμαι βουλευτή και είμαι και πρόεδρο και ε, δεν πάω να είμαι πρόεδρο, έχω και γνώμη όμω ω βουλευτή. Το έχω πει και στη διάσκεψη των προέδρων αυτό, των επιτροπών. Και ρώτησα και τον πρόεδρο Σούλτ τι πρέπει να κάνω. Ω πρόεδρο τη επιτροπή, ε, θα πρέπει στο βεστιάριο να αφήνω την προσωπική μου γνώμη. Και είπε ο κύριο Σούλτ, όχι βέβαια. Και ο κύριος Λάγκε ε, υπέστη επίθεση γιατί πήγε με τους σοσιαλιστές και δημοκράτες στην Ουάσιγκτον και να άκουσο ε, ε, τόλμησε να μιλήσει με τους Αμερικανούς όντας πρόεδρος Επιτροπής του Κοινοβουλίου. Εγώ τον υποστήριξα και ο πρόεδρος Σούλτς βεβαίω. Δηλαδή μπορεί να είσαι πρόεδρος αλλά δεν χάνεις την προσωπική σου γνώμη. Έχω το δικαίωμα να το κάνω, μόλις το έκανα. Ευχαριστώ για την κατανόηση. Το λόγο έχει τώρα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή Μάρκο Ντούρκο. Thank you, Chairman. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Δεν έχω να προσθέσω πολλά στην όλη συζήτηση, αλλά θα ήθελα να τονίσω παρόλα αυτά ένα δύο πράγματα. Ένα από τα ζητήματα τα οποία ετέθησαν αφορούσε την αεροπορία. Είχα πει και την προηγούμενη φορά ότι πράγματι θέτουμε τέτοια ζητήματα τα περιδιοκτησίας, για παράδειγμα, είναι ένα θέμα που το συζητούμε με τους Αμερικανούς συνομιλητές μας. Για το καμποτάζ. Εδώ τα πράγματα είναι λίγο ίσως πιο δύσκολα, διότι παραδοσιακά για λόγους όχι πάντα ευνόητους το καμποτάζ το πάντοτε από τις εμπορικές συμφωνίες. Δεν σημαίνει ότι πρέπει να είναι εντός, αλλά για το TTIP είναι ένα θέμα το καμποτάζ που στις εμπορικές συμφωνίες δεν συζητείται. Αυτό πρέπει να το έχουμε υπόψη. Όχι ότι θα πρέπει να ισχύσει το ίδιο και με την συμφωνία TTIP, αλλά δεν έχει γίνει σε αμυγός εμπορικέ συμφωνίες μέχρι τώρα. Νομίζω ότι αυτό είναι το μόνο που έχω να πω συγκεκριμένα για τα ζήματα που άπλονται το μέτρο μεταφορών και σα ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Ο εισηγητής για να κλείσει. Ευχαριστώ Πρόεδρε, σας ευχαριστώ πολύ. Κοιτάξτε, κατανοώ απολύτως και αντιλαμβάνομαι ότι η συμφωνία TTIP είναι πάρα πολύ επίμαχο θέμα και ε, πάρα πολύ συναισθηματικά φορτισμένο. Αλλά σας παραπέμπω στο εξή. Σήμερα σας έχω καταθέσει ένα κείμενο ως ένα πρώτο σχέδιο έχει αλλάξει από το πρώτο, από το αρχικό έτσι. Προσπαθήσαμε όσο γίνεται να βάλουμε στο συμβασμό όσες περισσότερες τροπολογίες μπορούσαμε. Την περασμένη Τετάρτη στο Στασβούργο κάναμε συμβαστικές τροπολογίες και προσπαθήσαμε και σας συστήλαμε σήμερα το πρωί. Εγώ χαίρομαι πάρα πολύ που λέγουν όλοι ότι είναι καλή γνωμοδότηση Και μετά, άμα θέλουν να την αλλάξουν 200%, τι θα μείνει από την αρχική γνωμοδότηση. Λέτε όλοι τι ωραία γνωμοδότηση και μετά αρχίζει το αλλά. Και θέλω να πω ότι ε, είναι κατέρωθεν απαραίτητη η ευελιξία. Και το λέω και προς τους συναδέλφους. Προσπάθησα να σημειώσω όλα τα σχόλια και τις παρατηρήσεις που ακούσαμε και σήμερα, αλλά δεν μπορώ να τα ενσωματώσω όλα, όπως καταλαβαίνετε. Διότι από τη μια έχω ε, ΕΛΚ, ΑΛΔΕ και συντηρητικούς, ε, οι τρεις αυτές ομάδες ε, είναι πιο συγκρατημένα θετική ας πούμε απέναντι στο TTIP αλλά έχω και τη συνάδελφο από την ΚΟΕ που είναι αναφανδόν κατά ε, και χρειάζεται πολύ μεγάλη τώρα πολιτική μαεστρία για να γράψεις μια γνωμοδότηση θα παραμείνω στην προσπάθεια αυτή θα τηρώ ενήμερους όλους τους και όδης ανεδεχτώ ενδεχομένως και άλλα κείμενα, αλλά θα πρέπει τελικά να καταλήξουμε σε μια ψηφοφορία. Υπάρχει διαδικασία και δεν μπορώ να τα βάλω όλοι. Εντάξει, να είμαστε προσεκτικοί απέναντι στο TTIP, να πούμε ξεκάθαρα ποια είναι τα θέματα των μεταφορών και τι πρέπει να προσεχθεί και από εκεί και πέρα πέμπτη πρωί ψηφίζουμε. Και στέλνουμε μια καλή γνωμοδότηση στην καθήλυνα αρμόδια επιτροπή. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ και για την εργασία και τη συνεργασία την τόσο αγαστή με τους σκιώδεις. Λοιπόν, στις μεταφορές θα ψηφίσουν την άλλη εβδομάδα, την 5η, 26 του μηνός Μαρτίου. Αυτό έχει προγραμματιστεί. Εντάξει, το ξέρουμε αυτό. Πάμε. στην Ίντα 6 και 7 Μαΐου και στην Ολομέλεια, στη δεύτε... Ε, μάλλον το Μάιο του 2015 στην Ολομέλεια. Αυτό είναι το χρονοδιάγραμμα, έτσι. Ωραία. Πάμε στο επόμενο θέμα στη μερίσια διάταξη. Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων και ε, τροποποίηση του προπολογισμού. Θα δώσω το λόγο πρώτα στους δύο εισηγητές, η Νέσα Γιάλα, Ladies First και μετά ο Ντομινίκη Ρικέ. Okay. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Εγώ νομίζω ότι ναι πράγματι μπορούμε να κάνουμε μια κοινή παρουσίαση διότι ήδη ο Ντομινίκ Ρικέ και εγώ δείξαμε ότι μπορούμε να εργαστούμε ομαδικά από κοινού και έτσι νομίζω ότι κερδίσαμε και την εμπιστοσύνη των μελών της Επιτροπής μας και για να προασπιστούμε και να διευρύνουμε το Connecting Europe Facility αλλά και να προωθήσουμε τα περί του ΕΣ αυτού του νέου Ταμείου Επενδύσεων. Θέλαμε να παραμείνει η διευκόλυνση μετά στην Ευρώπη το Connecting Europe Facility ως είχε μετά από μακρές διαπραγματεύσεις που κράτησαν χρόνια και ε, το Συμβούλιο, την πρόταση Κομισιόν, την πρόταση των κρατών μελών, των κλάδων, των περιφερειών, των εμπλεκόμενων. Όλα αυτά έπρεπε να τα μελετήσουμε και βήμα-βήμα. Πρώτα απ' όλα να βρούμε τα κριτήρια, μετά να δούμε τα έργα, τα σχέδια. Μέτρο-μέτρο προχωρήσαμε μέχρι το τελευταίο χιλιόμετρο, αν θέλετε, για να έχουμε μία πρόταση καλά καταρτισμένη και έχοντας ε, υπόψη μας και το πολύ πενιχρό προϋπολογισμό, πάλι Συμβούλιο, Κομισιόν, Κοινοβούλιο, νομίζω ότι καταφέραμε να καταλήξουμε στην άποψη ως πλειοψηφία ότι πρέπει να διατηρηθεί αυτό το μέσο. Γιατί θα πρέπει στην Ευρώπη να υπάρχουν και να βελτιωθούν όταν υπάρχουν οι υποδομές αυτές για να έχουμε και προστασία του περιβάλλοντος. Ήταν μεν μικρός ο προβλησμός, αλλά μπορούσαμε να ξεκινήσουμε να εργαζόμαστε με αυτό. Ξεκίνησε ο πρώτος διαγωνισμός, πάνε καλά τα πράγματα και είχαμε και μια καλή είδηση στη συνέχεια, το επενδυτικό σχέδιο του Juncker. Οποτε θα βελτιώσει και θα ε, δρομολογήσει την ανάπτυξη με βάση τι επενδύσεις. Αυτό μας βρίσκει σύμφωνος και το στηρίζουμε ως ιδέα. Βέβαια, ένα σχέδιο τέτοιο που έχει αυτή τη σημαντική συνιστόσα, τις επενδύσεις δηλαδή στις υποδομές, θα πρέπει να είναι συμπληρωματικό ή τέλο πάντων να αντλεί κάποια κονδύλια από το Connecting Europe Facility ή να γίνεται και το ανάποδο, αλλά όχι ένα σημαντικό κομμάτι του ΣΕΦ, του Connecting Europe Facility, να το ακροτηριάσουμε, να το κόψουμε και να το χρησιμοποιήσουμε για τις επενδύσεις ε, του σχεδίου Juncker. Διότι είναι σαν να έχουμε από το πρώτο διαγωνισμό ήδη καταδικάσει θάνατο αυτό το μηχανισμό, αυτή τη διευκόλυνση συνδέοντας την Ευρώπη. Υπάρχουν κάποιοι που έχουν υποβάλει προτάσεις αυτό το, στον πρώτο διαγωνισμό και άλλοι θα παρουσιάσουν προτάσεις σε άλλο, αλλά θα θεωρήσουν αυτοί που ήδη έχουν κάνει προτάσεις τους ότι εξαπατήθηκαν ή τέλος πάντων θα απογοητευθούν. Εμείς θέλουμε λοιπόν να διατηρήσουμε αφενός το ΣΕΦ και αφετέρου το ΕΦΣΥ το Ευρωπαϊκό Τεμιστατηγικών Επενδύσεων, τη νέα πρόταση, να ξεκινήσουμε ένα προπολογισμό Ξέρουμε ότι πάντα δυσκολευόμαστε να καταλήξουμε ο προλογισμό μεταξύ των τριών οργάνων. Αλλά ούτε η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων δεν θέλει ούτε εγγύηση ούτε μετρητά αυτή τη στιγμή. Υπάρχει και βέβαια και το θέμα της ευελιξίας. Θα μπορούσε αυτό να λειτουργήσει ως εγγύηση. Προσπαθούμε λοιπόν αυτό το σχέδιο έκθεσης να πούμε ότι απορρίπτουμε για τις επενδύσεις στις υποδομές και την εγγύηση που μας ζητάει η ΕΤΕ αυτά τα κονδύλια να βγουν από τον προπολογισμό του Connecting Europe Facility και προτείνουμε ως αντιστάθμιζα μα και συμφωνούμε με τους ε, συναδέλφους από την Επιτροπή Προπολογισμών και από την Επιτροπή Ήτρε ότι θα μπορούσαμε στα αποθεματικά ή με την ευελιξία, με το front loading, ε, την εμπροστοβαρή εκταμής κάποιων κονδυλίων, να μπορέσουμε να εξασφαλίσουμε αυτή την εγγύηση. Επίσης θέλαμε και στα ζητήματα της διακυβέρνησης θέλαμε να είναι και το Κοινοβούλιο ε, πρωταγωνιστής μαζί με τα άλλα θεσμικά όργανα, να είναι στην πρώτη γραμμή. Και επειδή θα ακολουθηθεί η κανονική διαδικασία κατά τη προπολογισμού και για το νέο Ευρωπαϊκό Ταμείο Στατικών Επενδύσεων, θέλουμε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο βάσει ακριβώ αυτή τη κανονική διαδικασία να συμμετέχει ισότιμα ευθύ εξ αρχή και από την Επιτροπή μας για τις μεταφορές δηλαδή θέλουμε να υπάρχει και ένα τομεακό κομμάτι σε, αυτή την, σε αυτό το ταμείο. Δηλαδή χρηματοδότες από την ΕΤΕ ή άλλοι επενδυτές που θα κάθονται στο τραπέζι για να πάρουν αποφάσεις. Σίγουρα είναι αυτοί οι οποίοι θα αποφασίζουν αν αυτό το προϊόν μπορεί να πουληθεί αλλά θα πρέπει να υπάρχουν και κάποιοι ειδικοί, κάποιοι προγνώσεις από τους διάφορους κλάδους. Και στην περίπτωσή μας, στην περίπτωση των μεταφορών, θέλουμε οι μεταφορές ε, να έχουν τον λιγότερο δυνατό κοινωνικονομικό αντίκτυπο. Και αυτά τα σχέδια θα πρέπει να τα προωθούμε λοιπόν. Έτσι θεωρούμε ότι θα πρέπει το πρόγραμμα Juncker να επηρεάσει επενδύσεις. Ε, στο άρθρο 5 λέμε ότι θα πρέπει να γίνει αυτά στο πλαίσιο της προσφοράς που θα προετοιμάσουμε με πάρα πολύ μεγάλη προσοχή για τα διευρωπαϊκά δίκτυα και τους διαδρόμους. Έχουμε το βασικό δίκτυο, έχουμε το παγκόσμιο δίκτυο. Σίγουρα δεν θα πρέπει να κάνουμε κανέναν περιορισμό γιατί υπήρχαν θα μπορούσαν οι εμπειρογνώμονες της ΕΤΕ να βρουν στα πλαίσια του βασικού δικτύου ή του παγκόσμιου τις ε, ευκαιρίες για να δημιουργήσουν εκεί επενδύσεις. Θα πρέπει απλά τα κριτήρια να είναι ευρωπαϊκά και για τα μελλοντικά δίκτυα, TEN, διευρωπαϊκά δίκτυα των μεταφορών. ως κίνητρο για τα κράτη-μέλη και επειδή υπάρχει μεγάλη φοδρόμηση και από το Συμβούλιο που είπε ότι θα βάλει ούτε ένα ευρώ στο Γενικό Ταμείο, τα κράτη-μέλη που χρειάζονται κίνητρα, παρακίνηση, ιδίω αυτά που, είναι, ε, που έχουν δυσκολίε ε, να εξεύουν σε χρηματοδότηση ή να κινδυνεύσουν αυτά τα δημόσια κονδύλια που θα χρειαστούν εμείς προωθούμε μια διαδικασία όπου οι επενδύσεις οι οποίες έχουν κοινωνικο-οικονομικό αντίκτυπο στο πλαίσιο του σχεδίου Juncker για τις υπηρεσίες στον τομέα των μεταφορών και τις σχετικές υποδομές θέλουμε να τηρούν τα κριτήρια του Συμφώνου Σταθερότητα. Σίγουρα ο Ντομινίκ θα μπορέσει να συμπληρώσει και να βελτιώσει αυτά που μόλι είπα. Ευχαριστώ. Πριν δώσω όμως το λόγο στον κύριο Ντομινίκ Ρικέ, θέλω να καλωσορίσω μια ομάδα επισκεπτών. Του κύριου Ρικέ έχουμε 20 φοιτητές. École Nationale des Ponts Καλωσορίσατε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Και είναι πάρα πολύ επίκαιρο τώρα ότι παίρνει το λόγο ο κύριος Ντομινίκ Ρικέ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα χαιρετήσω του τους φοιτητές που είναι και φοιτητές για τα θέματα των ε, συνδρομών. Εδώ ξεκινάει η ζωή ενός παλιού ζευγαριού που τα πάει και πολύ καλά, όπως είπε και ο συνάδελφος. Να ευχαριστήσω και τους σιώδους εισηγητές γιατί μερικά πράγματα πίεζαν τόσο πολύ που τους συναντήσαμε ήδη. Και ε, θα συμβάλλουν στην προετοιμασία της έκθεσης ώστε να έχουμε το μεγαλύτερο δυνατό βαθμό συμφωνίας και με εισηγητέ άλλων επιτροπών σε αυτή την περίπλοκη διαδικασία που προβλέπεται με τόσους πολλαπλούς εισηγητέ είχαμε συζητήσει πρόσφορες. Μπορέσαμε έτσι να φτάσουμε σε μια τοποθέτηση που δεν είναι απλώς αυτή της κάθε μιας επιτροπής ξεχωριστά, αλλά είναι η τοποθέτηση ολόκληρου του Κοινοβουλίου. Θεωρώ ότι είναι σημαντικό λοιπόν το Κοινοβούλιο να παραμείνει σταθερό στις θέσεις του το πρώτο που πρέπει να πω είναι κάτι που υπόθηκε. Ε, Βεβαίω στηρίζουμε την πρωτοβουλία να προβλεφθεί μια εγγύηση που να βασίζεται στο, ε, στα ευρωπαϊκά κονδύλια. Στον ευρωπαϊκό προπολογισμό μάλλον. Ε, μια εγγύηση που να αφορά τον εξοπλισμό την ε, συγκέντρωση μάλλον μακροπρόθεσμων επενδύσεων. Η απόρριψη κάποιων λύσεων μέσω του Connecting Europe Facility ε, ήταν κάτι που μέχρι τώρα δεν είχε πολύ νόημα. Εάν είμαστε σύμφωνοι με την πολιτική αρχή στην πράξη, όπως είπε και η θα πρέπει να κάνουμε κάποιες παρατηρήσεις. Το πρόβλημα του να εγγυηθεί κανείς έχει να κάνει με το κατά πόσον ε, διαθέτει ως εγγύηση, αυτό αποτελεί κείμενο της πρότασης της Επιτροπής, Κατά πόσον λοιπόν προβλέπει για αυτή την εγγύηση όσα προκύπτουν με τον καιρό λόγω των αναγκών. Το Ταμείο λοιπόν δεν θα πρέπει μόνο από το Connecting Group Facility και από το Horizon 2020 να πρεκοδοτηθούν, αλλά ακριβώς γιατί αυτά τα εργαλεία προβλέφθηκαν για να στηρίξουν μακροπόθεσμες επενδύσεις για τις υποδομές. Θα υπάρχει συνέπεια, αν γίνει κάτι τέτοιο και τα ερευνητικά προγράμματα που είναι δεύτερο πυλώνα των ε, ευρωπαϊκών επενδύσεων πρέπει να προστατευτούν. Είναι αποτελεσματικά, λειτουργούν καλά, δίνουν αποτελέσματα, έχουν συζητηθεί επιμακρών μεταξύ των διαφόρων συνόντων ε, στην Ευρωπαϊκή Ένωση μέχρι να αποφασιστούν και υπάρχουν και κάποια κρατικά προγράμματα, δημόσια προγράμματα μάλλον, που δικαιολογούνται μέσω αποδοτήσεων, όχι εγγύσεων, Υπό αυτέ τι προποθέσει λοιπόν ο μηχανισμό εγγύηση του Juncker δεν είναι ε, εύστοχο. Δηλαδή δεν θέλουμε να πάρουμε τα κονδύλια από ένα ταμείο, από ένα πρόγραμμα για να τα πάμε κάπου αλλού, να τα γδίσουμε για να ε, καλύψουμε άλλε ανάγκε. Θα ήταν κρίμα από την Ευρωπαϊκή Άποψη. Και έπειτα για την ε, διαδικασία του προπολογισμού με την εξαίρεση να μπορεί κανείς να πάρει τα κονδύλια που ε, ίσως να πλεονάζουν, αυτό δεν έχει νόημα εφόσον έχουμε μια διαδικασία τήσια με δύο βασικούς ε, υπεύθυνου να αποφασίζουν, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Για τους συναδέλφου λοιπόν τα λέω αυτά, κατά τη στιγμή που θα ετοιμάζουν τι τροπολογίε του, το θυμίζω ότι υπάρχει ανάγκη οι τροπολογίε σας να λαμβάνουν υπόψη τους κανόνες του αποπολογισμού. Το Ταμείο και η εγγύηση ε, καλύπτονται από το ε, ΑΑ του κανονισμού, του προπολογισμού. Όσοι δεν γνωρίζουν το κονδύλια από ένα στοιχείο του κανονισμού, του προπολογισμού, δεν μπορεί κανεί να πάρει κονδύλια από ένα ε, στοιχείο του προπολογισμού για να τα πάει καπάλου, Θα ήταν ιδιαίτερα περίπλοκη μετά τη διαδικασία και τελείωσε έκτακτη. Δεν μπορούμε να πάρουμε κονδύλια λόγου χάρη από κάποια ταμεία από το 1B ή το 4, το 5 και το 6 από τους τίτλους του προπολογισμού και να τα πάμε εκεί που θέλουμε, στο 1α λόγω χάρη. Οι τροπολογίες σας δεν θα γίνουν ε, αδεκτές από την περίπτωση. Από τεχνικής πλευράς. Έτσι, οι εισηγητές σας και οι εισηγητέ τη ΙΤΡΕ και είναι πολύ σημαντικό αυτό και για του εισηγητέ του Επιτροπή Προπολογισμών και τη ΕΚΟΝ που είναι επί τη ουσία υπεύθυνοι, πρότειναν να εξελιχθούν τα άρθρα 18 και 19 που ε, κυρίω προβλέπουν να λύσουμε από το Connecting Europe Facility και το Horizon 2020. Προτείνουν να ε, αντικατασταθούν από τις μη ε, προσδιορισμένες ε, υποχρεώσεις με την επιφύλαξη να πάρουμε από τα ειδικά ταμεία εφόσον υπάρξει απόλυτη ανάγκη. Όπως θα ξέρετε αυτό υπάρχει στον προπολογισμό, οι μη συγκεκριμένες, οι μη ε, προβλεπόμενες δεσμεύσεις. Εμείς, όπως ξέρατε, ε, είμαστε υπεύθυνοι για τα άρθρα 18, 19 και 5B. Ε, εκεί δεν θα επανέλθω. Χρειάζεται ένα σύστημα κυβέρνηση που να προστατεύσει τα συστήματα μεταφορών και τι υποδομέ βάσει των κατευθυντηρίων γραμμών, των διευρωπαϊκών δικτύων ε, και που να, προσ... να εξασφαλίζει την προστατευμένη ευρωπαϊκή αξία και όχι να είναι απλώς τραπεζικού χαρακτήρα και φύσης. Κατά τα άλλα, και για να μην επαναλάβω όσα υπόθηκαν, θα πρέπει να εκφραστούν ε, διαφορετικέ απόψει για την κυβέρνηση, για τον μηχανισμό που θέλουμε να προβλέψουμε εντό τη ΕΤΕ, για λόγου ταχύτητα και λειτουργικότητα και ελπίζουμε στον τραπεζικό αυτό μηχανισμό να ε, συμπεριλάβουμε στοιχεία ε, χρηστή πολιτική διακυβέρνηση, σωστή, η υπεύθυνη τη Ευρωπαϊκή Ένωση να προστατεύσουν όντω το ευρωπαϊκό συμφέρον και την ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία τους κινδύνους ούτως ή άλλως θα τους ε, καλύπτει η εγγύηση. Έτσι κι αλλιώς ο στόχο όλου του Ταμείου είναι η στήριξη των επενδύσεων. Να κλείσω λέγοντας ότι υπάρχει μια συγκεκριμένη θέση, σταθερή θέση του Κοινοβουλίου για την προέλευση των κονδυλίων της εγγύησης του Ταμείου, ότι πρέπει να σεβαστούμε τα όσα έχουμε δηλώσει, αλλά θα είναι ένα δύσκολο, δυσκερής γιατί θα πρέπει να διαφωνήσουμε και με το Συμβούλιο και με την Επιτροπή. Όπω ξέρετε, το όλο αυτό σχέδιο ε, εκπορεύεται απευθεία από τον ε, πρόεδρο Γιούνκερ. Θα πρέπει λοιπόν να μην ξεχνάμε και τον χρόνο που πιέζει, γιατί θα πρέπει λίγο να βιαστούμε και στα χρονοδιαγράμματα και στον τρόπο που δουλεύουμε. Πρόκειται για ένα κείμενο ιδιαίτερα σημαντικό και υπάρχει και μια διάσταση κατεξοχήν πολιτική αλλά και πολλά τεχνικά θέματα που δεν θα πρέπει να τα παραβλέπουμε γιατί έχουν και πολιτικές επιπτώσεις για το τι επιλογές θα κάνουμε. Για μένα είναι σαφές το Κοινοβούλιο πρέπει να παραμείνει συνασπισμένο, συσπηρωμένο στην ε, τυποθέτησή του. Διότι αν έχουμε σοβαρές αποκλήσεις θα βλάψουμε τις πολιτικές επιλογές που έχουμε προκρίνει όλοι μαζί εκ των προτέρων. Ευχαριστώ πολύ κύριε. Το λόγο έχει ο Μάρκος Πίπερ. Also ich Προσωπικά πιστεύω ότι για να βρεθεί ένα συμβιβασμός ε, μπορούμε από τώρα να καταθέσουμε διαφορετικέ απόψει, αλλά θα ήθελα ε, ρητά να ευχαριστήσω τους δύο για το πρώτο βήμα που κάναμε να σώσουμε κάπως το, τη διευκόλυνση συνδέοντας στην Ευρώπη, Connecting Europe. Όσο περισσότερα από τα αρχικά λεφτά σώσουμε, τόσο λιγότερο θα πρέπει να ανακατευθούμε με τα κριτήρια ε, στο σχέδιο του Juncker. Πιστεύω η επιλογή που έχει γίνει τώρα ότι είναι ένα πρώτο σημαντικό βήμα. Ως νέες πηγές χρηματοδότησης έχετε διαγράψει τις παραγράφους 18 και 19 που είμαστε πολύ υπέρ αυτού. Ε, ετήσια διαδικασία ζητάτε και λέτε ότι τα προγράμματα ε, από το 1α με περιθώρια, με το μέσο ευελιξίας κτλ. Και χρηματοδότηση ε, το πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο 16-20 θα πρέπει να επανεξεταστεί. Και όπου έχουμε ε, περίσευμα πλεόνασμα θα πρέπει να τα δίνουμε στο ΣΕΦ ή στην έρευνα. Όλα αυτά είναι ωραία και σωστά. Πλην όμως είναι αβέβαια. Ε, θεωρούνται, μάλλον δεν θα ε, ε, είναι αρκετά για να γίνουν δεκτά ως εγγύησεις. Πέντε email Μα στέλνουν οι επίτροποι τη μέρα και οι ίδιοι επίτροποι προτείνουν και τροπολογίε που θα του άρεσαν να βάλουν. Γιατί λένε δεν φτάνουν τα λεφτά αυτά για να είναι εγγύηση. Το καταλαβαίνω αυτό, διότι πρόκειται για ετήσια επανεξέταση, ενώ οι επενδύσει που θέλουμε εμεί να προκαλέσουμε ή να προσελκύσουμε είναι πολυετή. Αυτά δεν ασκούν ω εγγύηση, ε, ω ενέχειρο, ξέρω εγώ. Ε, αυτό που βρίσκω εγώ ενθαρρυντικό είναι ότι ούτε καν η ίδια Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, δεν αφισβητεί ότι ε, το Κοινοβούλιο θέλει οπωσδήποτε να διαγραφούν τα άρθρα 18 και 19. Είμαστε αποφασισμένοι. Και αν το καταλάβει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το χωνέψει και μας λέει ότι δεν περνάνε αυτά που ζητάτε εσείς, τότε ποιες είναι οι αρακτικές λύσεις αγαπητή Επίτροπη. Και μπαίνουμε εμείς τώρα στο παιχνίδι. Γιατί εμείς ως Κοινοβούλιο δεν έχουμε καν το δικαίωμα να ε, αλλάζουμε τις διατυπώσεις στον κανονισμό ή να κάνουμε συγκεκριμένες νομοθετικές προτάσεις. Δεν είναι δική μας δουλειά. Το μόνο που μπορούμε να κάνουμε είναι να καλέσουμε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ακόμα και να απαιτήσουμε να το κάνει για μας. Ε, θα πρέπει λοιπόν να δώσουμε μια εργαλειοθήκη ε, που να περιγράφουμε όσο γίνονται περισσότερα εργαλεία και συνειδητά λέω και από το 1β γιατί όχι, γιατί να μην το προτείνουμε, γιατί να μην το προσφέρουμε δεν βλάπτει τίποτα. Βοηθάει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να ε, το κοιτάξει. Εδώ είδαμε και ε, από την, στην αρμόδια επιτροπή ε, ε πώς μπορούμε να υποστηρίξουμε τα χρήματα στο ΣΕΦ, γιατί έχει και η Επιτροπή Μεταφορών. Να, κάνουμε μια προσφορά στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, μια εργαλειοθήκη, ότι ορίστε αυτές τις ιδέες σας προτείνουμε, βγάλτε κάτι λογικό από αυτά. Υποστηρίζω την προσέγγιση και της κυρίας Αγιάλα και του κυρίου Ρικέ, αλλά θέλω να τη συμπληρώσω και με άλλες ιδέες. Και παρακαλώ να υπερψηφίσει η Επιτροπή μας αυτό, γιατί εμείς ως Επιτροπή Μεταφορών έχουμε ένα καθήκον να αντιδράσουμε και να δράσουμε περισσότερο και από τους άλλους. Ο δεύτερος διαγωνισμός ε, σημαίνει ε, ότι το ΣΕΦ θα πεθάνει εκτός των χωρών συνοχής έχει βάλει και αρνητικά ποσά η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Καταλαβαίνετε ότι αν εξαιρεθούν οι χώρε συνοχή, έχει ταυτεί το πρόγραμμα. Αν δεν κάνουμε εμεί ό,τι μπορούμε, είναι δική μα δουλειά, το μεταφορών. Και ε, να βγούμε και λίγο από τα εσκαμμένα. Ε, χρειάζονται και άλλε ιδέε και ω Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα θα εργαστούμε προ την κατεύθυνση αυτή. Ένα τελευταίο σημείο. Για τα κριτήρια. Ε, δεν θα πρέπει να παραφορτώσουμε το σχέδιο του Γιούνκερ. Να μην ε, βάλει ό,τι θέλει το κοινοβούλιο. Ε, ακούω τα πιο τρελά πράγματα. Ε, γιατί και αυτό θα σημαίνει το θάνατο του σχεδίου Γιούνκερ. Τα κριτήρια ε, των διευρωπαϊκών δικτύων θα πρέπει να γίνουν σεβαστά, το κατανοούμε, αλλά να μην μπούμε σε υπερβολικές λεπτομέρειες γιατί θα παραφορτώσουμε το σχέδιο αυτό και θα μπλοκάρουμε και τη διαδικασία της Ευρωπαϊκής Τράπεζας επένδυσης που έχει τον πρώτο λόγο. Ε, δηλαδή, ε, επί ξηρού αχμής βρισκόμαστε και ε, ε, όσο σεβόμαστε και σώζουμε το Connecting Europe, τόσο λιγότερο αναμειγνυόμαστε και μπαίνουμε στα πόδια του Juncker με το σχέδιό του. Ευχαριστώ. Η κυρία Τζάκη Φώστερ. Thank you, um, Chairman. Thank you to the... Ευχαριστώ Πρόεδρε, ευχαριστώ και τους εισηγητές. Έχω από τον κύριο Σίλε, τον σχεδόν εισηγητή μας, μια, ένα σημείωμα και θα σας διαβάσω. Τι έγραψε. Στα λετωνικά. Στα λετωνικά, ναι, ναι, στα λετωνικά. Νομίζω μάλλον θα μείνω στα αγγλικά, είναι καλύτερα τα λετωνικά. Ο κ. λέει για του εισηγητέ, οι βασικέ του παρατηρήσει είναι ότι το ταμείο αυτό θα πρέπει να είναι προσωρινό όχημα. Οι συντηρητικοί και μεταρρυθμιστέ πιστεύουν ότι το ταμείο αυτό αρχικά προβλέφθηκε ω προσωρινή λύση για να ε, αντιμετωπίσουμε τον αρνητικό κύκλο επενδύσεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ανησυχούμε ωστόσο ότι η πρόταση για το ΕΦΣΥ έχει σκοπό να το προβλέψει ω ένα διαρκέ μέσο. Επίση, προβλέπεται να διευκολύνει την υλοποίηση ασφαλέστερων και προσανατολισμένο προ τι επιχειρήσει αλλά και βιωσιμότερων ε, προγραμμάτων για τι υποδομέ των μεταφορών με μεγάλο κέρδο. Ιδίω τα βιομηχανικά κέντρα. Σε αυτέ τι περιπτώσει, χωρί συνοριακέ διασυνδέσει, αυτό δεν θα λειτουργήσει. Οι στόχοι όμω του, του Connecting Europe Facility και των διευρωπαϊκών δικτύων ε, προβλέπουν τόσο άλλω διασυνοριακά προγράμματα κοινού συμφέροντο που συνήθω λειτουργούν με χαμηλό κέρδο. Άρα ε, οι συντηρητικοί και μεταρρυθμιστέ καλωσορίζουν την ξεκάθαρη διασύνδεση σύνδεση ε, του ΕΨΙ με το Connecting Europe Facility και το TNT αλλά και τους ε, κανονισμούς τους. Θα αλλάξει η βασική φιλοσοφία βεβαίω τη πολιτική για τα διευρωπαϊκά δίκτυα εφόσον χρησιμοποιηθεί το ΕΦΣΥ και θα πρέπει να δούμε τι θα γίνει με την ελληνική και τη συνοχή. Τέλο, ό,τι αφορά τη χρηματοδότηση, εκ πρώτη όψη μπορεί να φαίνεται μια καλή λύση να μην αγγίξουμε τα χαρτοφυλάκια του Horizon 2020 και το C, το Connected Europe Facility για να χρηματοδοτήσουμε το EFSI, αλλά ο κ. Σίλερ έχει και εναλλακτικέ προτάσει να χρηματοδοτηθεί το EFSI από τον επαναπρογραμματισμό κοντιλίων εντό του Ευρωπαϊκού Προπολογισμού ετησίω. Αυτό είναι κρίσιμη σημασία για την λήψη αποφάσεων, αλλά έτσι θα μπορέσει να γίνει και η ανακατανομή των πλεονάζοντων κοντιλίων πιο προβλέψιμη. Στου τίτλου 1α του ε, πολιτικού το δημοσιονομικού πλαισίου και από το ε, Ταμείο των Επιδόσεων από τη Γεωργία και τα Διευθυντικά Ταμεία, από το 1Β δηλαδή, θα μπορούσαμε να πάρουμε επιπλέον κονδύλια. Αυτά είναι τα σχόλια του κ. Σίλερ και αν χρειάζονται διευκρινήσει ε, ο οι εισηγητέ μάλλον. Οι, οι συνεισηγητέ ευχαρίστω να τι λάβουν από τον Ρόμπερτ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ, κύριε Μάισνερ. Ναι, Ευχαριστώ δεν έχω τόσα πολλά να προσθέσω κι εγώ. Οι συγητέ τα ξέρουν πολύ καλά και πραγματικά είναι ένα παλιό ζευγάρι σε αυτά τα θέματα τα δημοσιονομικά. Αυτό τώρα είναι φιλοφρόνηση ή όχι, λέει ο Πρόεδρο. Μα το είπε ο ίδιο ο κύριο Ρικέ. Εγώ το επαναλαμβάνω, δεν κάνω τίποτα παραπάνω. Ε, η μεγάλη δυσκολία για μα ποια είναι. Ότι τα λεφτά θα τα πάρουν από τι μεταφορέ. Εντάξει, Ντομινίκ, θα τα βρούμε μεταξύ μα. Ε, ε, να με συμπαθά. Λοιπόν, ε, από το Connecting Europe θέλουν να τα πάρουν τα λεφτά, αυτό είναι το θέμα και εμείς δεν το θέλουμε. Περί αυτού πρόκειται. Πολλά υπόθηκαν σωστά, να μην είναι πάρα πολύ στενά τα κριτήρια, είπε ο Πίπερ, αλλιώς θα παραφορτώσει το σχέδιο Juncker, ε, που το θέλουμε, δεν θέλουμε να αναβαγίσει, αλλά το θέμα είναι πόθεν θα βρεθούν τα λεφτά. Και ε, συμφωνώ απολύτως με αυτά που είπαν οι δύο εισηγητές μας τώρα ότι θα πρέπει το 18 και το 19 άρθρο να μην περάσουν όπως έχουν, δηλαδή από τα υπόλοιπα ε, και τα πλεονάσματα που έχουν, ε, αλλά εμείς πώς θα πείσουμε τα κράτη-μέλη όταν περισσεύουν κάποια λεφτά να μην τα ζητάνε πίσω, αλλά να τα δίνουν για την Ευρώπη, που πραγματικά θα σημάνει ανάπτυξη. Ε, στη θεωρία το σχέδιο Γιούνκερ είναι πολύ ωραίο και το υποστηρίζω απολύτω. Και ε, όταν είσαι ιδιώτης επενδυτής χρειάζεσαι κίνητρα. Πώς μπορούμε να τους προσελκύσουμε. Δεν θέλουν και αυτοί να είναι πολύ στενός ο κορσές για να επενδύσουν. Αυτό πώς θα το πετύχουμε όμως ε, χωρίς να χάσουμε τα χρήματα του ΣΕΦ που, που φτύσαμε αίμα για να τα πετύχουμε. Δεν μπορούμε να τα βάλουμε αυτά ως ε, ασφάλεια, ως εγγύηση. Κάπως Είμαστε τώρα σε ένα φαύλο κύκλο και ψάχνουμε μια στρατηγική για να βγούμε από αυτό το αδιέξοδο. Έχετε καμιά ιδέα πώς να πείσουμε τα κράτη-μέλη να μην τους επανακαταβάλλονται τα που ε, απομένουν, αλλά να δοθούν για ένα κοινό ευρωπαϊκό σκοπό. Θα ήταν μια πολύ καλή ευρωπαϊκή παραλλαγή αυτή. Θα το πετύχουμε από φέτος. Και από άλλες πηγές, αν αρχίσουμε ήδη από φέτος να ξυλώνουμε ε, άλλα λεφτά, ποια είναι αυτά. Ή θα είναι πάλι το ΣΕΦ και ορίζον 2020. Αλλά τότε θα έχουμε ήδη υποπέσει στο πρώτο ε, αμάρτημα. Δεν ξέρω πώς το βλέπουν οι υπόλοιποι σκεδοσυγητές, αλλά όλοι γι' αυτό μιλάνε. Ευχαριστώ. Η κυρία Κίλωνεν. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Προς τους εισηγητές να πω ότι τους ευχαριστώ για την ε, ομαδική τους δουλειά. Αυτό που δεικνύει ότι η Επιτροπή μας είναι έτοιμη να αγωνιστεί για, την, για το σκέλος της χρηματοδότησης. Υπάρχουν κάποιες επαναστατικές ιδέες. φρόντισαν να τις θέσω σε, αυτή την, σε αυτόν τον ε, κοινό αγώνα και στην Φινλανδία γνωρίζουμε πολύ καλά και το τι θα πει αγώνα και το τι θα πει κονδύλια. Οπότε, το ζήτημα είναι κατά πόσο να έχουμε όλα τα μέσα στη διάθεσή μας για να αγωνιστούμε για τα χρήματα που επιζητούμε να έχουμε και αν θα παραμείνουμε πιστοί στους πολύ καλούς στόχους που έχουν θέσει οι συνεισηγητές. Εάν δείτε τις υποδομές που έχουμε τώρα, και τους στόχους του προπολογισμού, αλλά και το τι στόχους θέλουμε να πετύχουμε για τι μεταφορές, το ερώτημα είναι κατά πόσο μπορούμε να προσφέρουμε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή κάτι καινούριο. Μια νέα φιλοσοφία που θα επιτρέψει να ε, υπάρξει πρόοδος στην απασχόληση και την ανάπτυξη, κάτι που θα αρέσει και στους επενδυτές διότι στον τομέα των μεταφορών τα τελευταία χρόνια Όταν ε, τελείωναν τα κονδύλια, ε, κάποιες μας καταφέρναμε όλα αυτά καλά αποτελέσματα. Αν και βέβαια πρέπει κανείς να βρει μια ε, άλλη λύση στην πολιτική. η αγάπη μόνη της δεν αρκεί, δεν κάνει κανένα τίποτα από αγάπη, αν και πολλές φορές χρησιμεύει για να συνδυάσει τα πράγματα. Τώρα για τη διασύνδεση των μεταφορών με την ενέργεια. Πρέπει και αυτή την ιδέα να την προάγουμε, ώστε οι ευθείες μεταφορές, ο προγραμματισμός των μεταφορών, η διαλογικότητα των μέσων μεταφοράς και η συμμετοχή όλης της κοινωνίας είναι στόχοι που θέλουμε να πετύχουμε. Πρέπει να τα περιγράψουμε σωστά ώστε τα υπάρχοντα κονδύλια να τα αξιοποιήσουμε με πιο έξυπνο τρόπο και να διατεθούν στο ευρωπαϊκό σύστημα μεταφορών. Το ερώτημα είναι πώς μπορούμε να αποδείξουμε ότι οι σιδηρόδρομοι, οι λιμένες, τα αεροδρόμια, οι αυτοκινητόδρομοι δεν θα ε, κατασκευαστούν ως αυτός σκοπός, αλλά ότι θα έχουν πρόθεση να ε, διευκολύνουν τους πολίτες της Ευρώπης, να ε, προσφέρουν υπηρεσίες μεταφορών, να στηρίξουν το σύστημα μεταφορών στην Ευρώπη. Πώς θα προσελκύσουμε λοιπόν επενδυτές στο σύστημα μεταφορών αν δεν προσφέρουμε ένα τέτοιο σύστημα όπου οι προκλήσεις της διοργάνωσης, της διαχείρισης του κυκλοφορικού η πρακτική διοργάνωση των υπηρεσιών δημόσιας μεταφοράς, η προσέγγιση, η φιλική προς τον πελάτη, αλλά και η τεχνογνωσία για τον τομέα συνολικά δεν υπάρχουν. Αυτά πρέπει να φέρουμε ε, στη συζήτηση για να μπορέσουμε να προασπιστούμε το ε, πρότυπο χρηματοδότησης του Connecting Europe Facility. Και τα λέω όλα αυτά διότι πρέπει να είμαστε σβέλτοι και να έχουμε και ένα εναλλακτικό σενάριο ή πλάνο. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα φέρει πολλές αντιρρήσεις και πιστεύω ότι θα είναι αρκετά αμετακίνητη. Είμαι λοιπόν κάπως ίσως η ευρωπαικη επιτροπη θα φερει πολλες αντιρρησεις και πιστευω οτι θα ειναι τα αμετακινητη ειμαι λοιπον καπως ισως η παλακιδα του ζευγαριού αυτού που εργάζεται πριν της Σας ευχαριστούμε κυρία Ντελή. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θέλω να ευχαριστήσω τους ε, συνεισηγητές για τη δουλειά τους. Νομίζω ότι δικαιούμαστε ως Επιτροπή και ως Κοινοβούλιο, δικαιούμαστε λοιπόν να θέσουμε το εξή πρώτο ερώτημα για το σχέδιο Juncker. Πολύ απλά, ποιος θα διαλέξει τα προσχρηματοδότηση έργα. Και ακριβώς ε, στο Ταμείο Σταδικών Επενδύσεων γνωρίζουμε ότι σήμερα υπάρχει ένα εποπτικό συμβούλιο που ε, εκπροσωπούνται εκεί η ΕΤΕ, η Κομισιόν, αυτοί δηλαδή που θα ορίσουν τις προτεραιότητες, τις στρατικές προτεραιότητες και τις γενικές κατευθύνσεις. Εγώ θέλω να σας πω ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι μία από τις δύο αρχές επί του προπολογισμού. Εμέσως λοιπόν ε, συμβάλλει και αυτό όπως και η ΕΤΕ και, το, και η Κομισιόν. Επομένως είναι απόλυτα θεμητό να απαιτήσει να εκπροσωπείται σε αυτό το οπτικό Συμβούλιο για την επιλογή των διαφόρων έργων και προγραμμάτων. Υπενθυμίζω ότι η τοπική αυτοδιοίκηση ε, ε, κλείστηκε από τον όλο Είναι καλό αυτό το μήνυμα που δίνουμε Έχουμε μία, ένα μήνυμα από τα πάνω προς τα κάτω. Εμείς όμως θέλουμε να ζει στις περιφέρειες ε, και να ε, ανεβαίνει από κάτω προς τα πάνω, όχι το ανάποδο. Εμείς οικολόγοι θέλουμε να προτείνουμε διαφοροποιήσεις στις δύο προτάσεις. Καταρχάς, άρθρο 5, ξεκάθαρα θέλουμε εκεί να αναφέρονται τα βασικά κριτήρια και οι προϋποθέσεις χρηματοδότησης σχεδίων στο δεμέτρο μεταφορών. Όπως έγινε στο ΕΜΙΕ. Το e βλέπαμε στα δυσνοριακά πώ ελαστικοποιεί το εξωτερικό κόστο, μειώνονται οι εκπομπέ του του άνθρακα, ε, γίνονται σεβαστοί οι περιβαλλοντικοί κανόνε κτλ. κτλ. Επίση, θα καταθέσουμε τροπολογίες για να υπογραμμίσουμε τη σημασία να υπάρχουν συνέργειες μεταξύ μεταφορών τηλεπικοινωνιών και ενεργειακών δικτύων, όπως λέγεται στον κανονισμό. Όπω e Όπως και στο RTMS ε, για τη σήμα, σηματοδότηση, για τους σιδηροδρόμους ή το EST. Τα ευφύ δίκτυα μεταφορών και τα συστήματα ε, πληροφοριών ε, για τις ε, πλωτές μεταφορές. Επίσης, έχουμε το θέμα της συγχωρήπανσης των συνδρομικών μεταφορών. Προτείνουμε επίσης χρηματοδότηση ως προτεραιότητα των περιφερειακών και συνοριακών συνδρομικών δικτύων που λείπουν, που εγκαταλείφθηκαν εντελώς ή διαλύθηκαν και για τις υποδομές, ε, για τους ποδηλάτες. Επίσης, 19. Θέλουμε να διαγραφεί αυτό το άρθρο, το προτείνει και το σχέδιο της γνωμοδότησης, το ή άλλως. Και τέλος, θα καταθέσουμε τροπολογίες σε σχέση με αυτό που είπα, σε ό,τι αφορά το σχέδιο προπολογισμού υπαρθμών 1 και για το γενικό προπολογισμό του 2015. Ευχαριστώ. Rosa D'Amato. Ευχαριστώ, η Ματ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Είμαστε ιδιαίτερα ικανοποιημένοι με τι κοινέ θέσει, όπω διατυπώθηκαν. Η διαγραφή των άρθρων 18 και 19 μέσα του σύμφωνου. Η πρόταση τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή να χρηματοδοτήσει ένα σημαντικό μέρο ε, του Ταμείου από το Horizon 2020 και του Connecting Europe Facility δεν μα πείθει καθόλου. Μάλιστα, ε, επιβαρύνει πάρα πολύ τους τομείς για τους οποίους οι υποδομές με δυσκολία προσελκύουν τα ιδιωτικά κεφάλαια. 8 δις που ε, μεταξύ ε, που προέρχονται στο ΕΦΣΥ, 3,3 προέρχονται από το Connecting Europe Facility και μόνο 2 θα κατευθυνθούν στις μεταφορές. Η, τα κονδύλια του Connecting Group Facility γίνονται τελικά ως ε, επιδοτήσεις μαζί με τα κονδύλια των 100 μελών, χρηματοδοτούν συστήματα μεταφορών που ε, δύσκολα θα καλύπτονταν από τις θετικές επενδύσεις. Κάτι που προβλέπει ο κανονισμός ΕΨΗ μεταξύ των 2,8 δις, κάποια ε, στι στις οδικές και συντοματικές ε, διασυνδέσεις ε, που ουσιαστικά δεν φέρνουν μεγάλο κέρδος. Αυτό ε, θα δημιουργήσει δυσκολίες στην έννοια των τεχνολογιών και στην προσελκύση ιδιωτικών κεφαλαίων. Ακόμη και με μικρότερο πολλαπλασιαστή από αυτόν που έχει υπολογιστή για τη μόχλευση του 1 προς 15. Εδώ λοιπόν κάποια πράγματα θα θέλαμε να τα συζητήσουμε με τους συζητητές, όπως για παράδειγμα τη διάθεση να επιτύχουμε ακόμη και ε, με τρόπο που θέσει ε, χρηματοδότηση από το κεφάλαιο 1α ε, για την αναπτύξη και την απασχόληση, ιδίω σε περίοδου λιτότητα όπω αυτή η περίπτωση που ζούμε. Θα πρέπει επίση μαζί με του ε, συντονιστέ να μελετήσουμε την αιτήσια κατανομή του προπολογισμού. Δηλαδή, δεδομένου ότι το ΕΦΣΥ μπορεί να γίνει ίδιο πόρο για να καταπολεμήσουμε την ανητυχία, για να ξεπεράσουμε αυτή την κρίση, τότε θα πρέπει το Ταμείο αυτό να λειτουργήσει πληρωματικά. Οπότε διερωτώμαστε μήπως αυτή η ετήσια ε, ανακατανομή γίνει ε, μια επιπλέον τροχοπέδη που θα φέρει ε, τις εγγύσεις που θα θέλαμε να έχουμε και αποδυναμώνει την όλη προσπάθεια. Ελπίζουμε να μπορέσουμε να συνεργαστούμε για τις δύο αυτές προτεραιότητες. Η Ρεβονταλόν. Ένα μεγάλο ευχαριστώ για τη δουλειά και των δύο συνεισηγητών που επέλεξαν να ακολουθήσουν μια οικοδομητική συλλογική προσέγγιση και να μην είναι τομεακή προσέγγιση και ο καθένας να υποστηρίζει τα του οίκου του. Αυτό το σχέδιο δείχνει ότι αν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι ενωμένο, αν ε, οι επιτροπές θελήσουν ε, να προσπίσουν από κοινού τα συμφέροντα του Κοινοβουλίου μπορούμε να μετακινήσουμε κάποιους που έχουν να απόψει απόψεις ό,τι αφορά τη, το διευκόλυνση στην Ευρώπη ή τον ορίζοντα 2020 που θα χρηματοδοτήσει το Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων. Οι μεταφορές, η ανάπτυξη των ευρωπαϊκών δικτύων που έχουν προστέμενη ευρωπαϊκή αξία πρέπει να είναι αναπόσπαστο τμήμα των δυνατοτήτων χρηματοδότηση του Ταμείου Στρατηγικών Επενδύσεων. Αριθμιστικά τώρα έχουν τροπολογία 41. Προτείνει διεύρυνση τη επενδύσεων για να αποκλείεται από τον υπολογισμό του ελλείμματο ε, ο προϋπολογισμός των σχεδίων που θα χρηματοδοτηθούν από αυτό το Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων. Αυτό θα βοηθήσει να ανακάμψουν δημόσιες επενδύσεις. Ε, πρέπει επίση να τονίσουμε τι προτάσει τη κοινή έκθεση Econ Budget για την υλοποίηση του Ταμείου Στατικών Επενδύσεων που βελτιώνει το κύμα της Κομισιόν. Σε ό,τι αφορά τη διακυβέρνηση πρώτα απ' όλα, δίνει τη δυνατότητα στους βουλευτές να είναι σε αυτή τη, το Εποπτικό Συμβούλιο, άρα ε, να επηρεάζουν και για τον ορισμό του Γενικού Διευθυντή, για την υπογραφή της συμφωνίας μεταξύ Κομισιών ΕΤΕ. Στέλνουμε λοιπόν έτσι ένα ηχηρό μήνυμα ότι το Κοινοβούλιο που εκπροσωπεί τη Φωνή των Ευρωπαίων Πολιτών πρέπει να γνωμοδοτεί στο πλαίσιο ε, του Ταμείου Στρατηγικών Επενδύσεων και για την επιλογή των έργων. Έχουμε τα προσθετικότητας. Ε, θα βελτιώσει την προσθέμενη αξία του Ταμείου το Κοινοβούλιο αν εξασφαλίσει ότι θα πηγαίνουν σε έργα με πραγματική ευρωπαϊκή προσθέμενη αξία που δεν θα τα χρηματοδοτούσε η ε, ΕΤΕ αυτά τα κονδύλια. Ευχαριστώ. Ε, Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Όλοι είναι υπέρ του ταμείου αυτού, του ΕΦΣΙ, του Ταμείου Στρατηγικών Επενδύσεων. Αλλά όλοι θέλουν να ρίξουν 315 δισεκατομμύρια στην ευρωπαϊκή οικονομία, αλλά ας είμαστε ειλικρινείς. Διαβάζοντας την έκθεση των δύο συνεισηγητών μας, τότε είναι μεγάλη πρόκληση να δώσουμε σάρκα και οστά σε αυτό το ταμείο. Είναι τεράστια πρόκληση και το λέω θετικά. Θα μπορούσα να το πω και μέγα πρόβλημα. Με ενδιαφέρον σημείωσα την έκθεση αυτή, ιδιαίτερα την εισαγωγή στην εισαγωγή τους, ε, εκ των προτέρων δηλαδή, βάζουν κάποια πολιτικά σημεία οι εισηγητές και με οξύ τρόπο για το τι θέλουν και ποια θα είναι η δική μας συνεισφορά, της Επιτροπής Μεταφορών εννοώ, και συμφωνώ με αυτά. Και σας εύχομαι πολύ μεγάλη επιτυχία στις διαπραγματεύσεις, γιατί εκεί θα είναι πολύ περίπλοκα τα πράγματα από αυτά που ακούω σε διάφορες φήμες στον διαδρόμο, τι μπορεί και τι δεν μπορεί να περάσει και τι επιτρέπεται και τι όχι. Πρόεδρε, εμείς ως Επιτροπή Μεταφορών έχουμε τεράστιο πρόβλημα με τη χρηματοδότηση ε, του Ταμείου Στρατηγικών Επενδύσεων. Έχει κατατεθεί μια πρόταση, άρθρα 18 και 19 να διαγραφούν, αλλά ως καλό κοινοβούλιο θα πρέπει να φέρουμε και εναλλακτικέ προτάσεις όταν λέμε κάτι να σβήσουμε και ο συνάδελφος Μάρκους Πίπερ ήδη πρότεινε μια εργαλειοθήκη να φέρουμε ε, με διάφορα ισοδύναμα και εναλλακτικά για τη χρηματοδότηση. Εγώ μπορώ να σας πω εξ ονόματος του ΕΛΚ ότι εμείς είμαστε υπέρ της διεύρυνσης της χρηματοδότησης. Οι συνάδελφοί μου έχουν γράψει μια επιστολή, μάλλον να το πω αλλιώς, έτσι τους προβληματίζει, αλλά δεν επιτρέπεται να πάρουν τα λεφτά μόνο από το ΣΕΦ και το ορίζοντα 2020 και τα περιθώρια του γενικού προπολογισμού και τα περιθώρια στη συνοχή να μην αξιοποιούνται. Είναι τρελό αυτό. Και είναι καλό η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να κοιτάξει τη διεύρυνση της χρηματοδότησης και να καταλάβει ότι θα είναι και κόκκινη γραμμή για το Κοινοβούλιο. Δεύτερο, το περίγραψε πολύ καλά η κυρία Γιάλα Σέντερ. Με το ΣΕΦ και τα διευρωπαϊκά δίκτυα περίγραψε πολύ καλά τα έργα. Και εμείς ως Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θέλουμε στην τράπεζα επενδύσεων, δεν ξέρω πώς γίνεται καλά steering committee, project line, δεν ξέρω πώς τα λένε, να επηρεάζουμε πάντως στην Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων τα έργα που θα επιλέγονται. Δεν επιτρέπεται να απεμβολήσουμε όλα τα λεφτά από την ε, συνδέοντα στην Ευρώπη και να πάει, ξέρω εγώ, όλο αυτό το, το χρήμα στην ε, ε βιομηχανία στον κλάδο του διαδικτύου. Ξέρω ότι ανήκουμε ε, στην ίδια σχολή σκέψης θέλουμε και χρήματα για τα κλασικά έργα υποδομής. Εσωτερικές σε πλωτές οδούς και σε δυρόδρομο Και θα πρέπει να έχουν θέση στο ταμείο αυτό. Γιατί είναι πάρα πολύ σύγχρονο και μοντέρνο να τα βάζουμε όλα στα κομπιούτερ και στα ε, συστήματα διοδίων σούπερ ε, που να είναι ψηφιακά. Αλλά εμείς Είμαστε υπεύθυνοι για τις κλασικές υποδομές, για τις συνδυασμένες μεταφορές, για το σιδηρόδρομο και τις εσωτερικές πλωτές οδούς. Συνοψίζω. Ευρύτερη χρηματοδότηση. Περισσότερη επιρροή και λόγο να έχει το Κοινοβούλιο για την επιλογή των έργων της ε, ΕΤΕ και προσοχή στα κλασικά έργα υποδομής. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Ισμαήλ Αρτούκ. Ευχαριστώ και όλους του συζητητέ και τους κοιόδη ε, από ε, τις διάφορες πολιτικές ομάδες και τις εισηγήτριες. Κοιτάξτε, υπόθηκαν ήδη πολλά, ε, με τα οποία συμφωνώ. Θέλω να τονίσω μόνο κάτι. Που μέχρι τώρα μόνο η Καϊρημάντελή το είπε τι θα κάνουμε και τι θέλουμε να κάνουμε με την επιλογή των έργων. Και ο συνάδελφος Πίπερ και άλλοι είπαν τι δεν επιτρέπεται, ε, συμφωνώ απολύτως, Πριν όμως πρέπει να δούμε και τι θα επιτρέπεται. Και δεν επιτρέπεται το ευρωπαϊκό επίπεδο να γίνεται ρήμην του Κοινοβουλίου. Κάπως θα πρέπει να χρηματοδοτήσουμε κι εμείς σε ευρωπαϊκό επίπεδο, δεν διαφωνούμε. Αλλά για να γίνει αυτό θα πρέπει το Κοινοβούλιο, αν όχι η Επιτροπή μας, να μπορεί να αποφασίζει ποια έργα επιλέγονται με βάση ποια κριτήρια. Όλη αυτή η δουλειά μπορεί κανείς, ας πούμε το, από το Συμβούλιο, ή από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να την αντιμετωπίσει βάζοντας κριτήρια. Εμείς δεν θα πρέπει να επανεφεύρουμε το τροχό. Την τελευταία περίοδο έχουμε συζητήσει τι θέλουμε να κάνουμε με το χρηματοδοτικό μηχανισμό διασυνέοντας στην Ευρώπη και ποιες είναι οι κατευθυντήριες γραμμές των ε, διευρωπαϊκών δικτύων μεταφορών. Τόσο χρόνο χρειαστήκαμε για να ορίσουμε κριτήρια σαφή και στραμμένα προς το μέλλον που μπορούν να εφαρμοστούν και θα έπρεπε και στο Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων. Δεν χρειάζεται να επανεφεύρουμε τον τροχό, επαναλαμβάνω. Τον έχουμε βρει και σε αυτό το steering committee ε, θα πρέπει να συμμετέχει και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο κάπως να λαμβάνεται υπόψη. Θα βρούμε με ποιο τρόπο, ποιος και πώς θα μας εκπροσωπεί ως Κοινοβούλιο. Αλλά ότι κάποιο λόγο πρέπει να έχουμε και εμείς είναι νομίζω αδιαφυσβήτητο. Τελευταίο θέμα. Είναι πάρα κινδυνευμένο και τυχοδιοκτικό θα έλεγα αυτό όχι από τη σκοπιά της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αλλά του Συμβουλίου. ότι δεν συμμετέχει καν στη χρηματοδότηση αφενός καφετέρου με ίσχυτη τη συνείδηση, το είπαν και οι Υπουργοί Μεταφορών ή δεν ξέρω, μάλιστα αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων, το Συμβούλιο που πέρασε άρον-άρον το σχέδιο Juncker, αλλά κανείς και καμία από τους πρωθυπουργού δεν μπήκε στον κόπο να ρωτήσει πού θα βρουν τα λεφτά. Τα έχετε πάρει από πού, έχουν σημασία για κάποιο άλλο, τι κονδύλια είναι αυτά, υπάρχει η ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία, τους ήταν μάλλον αδιάφορο. Ε, έχουμε την εντύπωση ότι θέλουν να το διεκπαιρεώσουν κακήν κακός, αλλά θα πρέπει να επιτρέπεται να τους ρωτήσουμε πώς είναι δυνατόν ε, έτσι ελαφρά την καρδία και χωρίς μεγάλες αντιστάσεις να επιτρέψουν ε, λεφτά από υποδομές, έρευνα, ανάπτυξη, ευρυζωνικότητα, ενέργεια, έτσι χωρίς να συμμετέχουν καθόλου τα κράτη-μέλη στην απόφαση αυτή. Τελευταίο, δεν επιτρέπεται, επαναλαμβάνω, τα κράτη-μέλη να είναι και οι μεγάλοι κερδισμένοι. Καλά, ποιο άλλο δεν θα είναι. Διότι αν απογειωθεί αυτό το σχέδιο Juncker, αν αρχίσει να λειτουργεί, είναι προ όφελος των κρατών μελών. Έτσι δεν είναι. Οπότε το ελάχιστο θα είναι να συμμετέχουν και στη χρηματοδότηση και το Κοινοβούλιο ε, βεβαίως να έχει λόγο και για την επιλογή των έργων. Ευχαριστώ. Ο κύριος Κούν. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Σημαντικό είναι που συμφωνούμε τουλάχιστον καταρχήν ότι τα χρήματα που δίνει η Ευρωπαϊκή Ένωση για τις υποδομές και για τις μεταφορές θα πρέπει να παραμένουν σε αυτό τον κορβανά. Άρα οι δύο παράγραφοι άρθρα 18 και 19 θα πρέπει να διαγραφούν και σε καμία περίπτωση να μην τεθούν σε ισχύ. Θα έκανα όμως μια άλλη πρόταση εγώ. Από το ΣΕΦ και τους διαδρόμους των διευρωπαϊκών δικτύων θα πρέπει να βγάλουμε όλα τα μεγάλα έργα που δεν μπορούν να χρηματοδοτηθούν από εκεί. Γιατί αυτές είναι οι δυνατότητες για το επενδυτικό σχέδιο και το ταμείο που μπορεί να εφαρμοστεί στην πράξη. Αν κοιτάξουμε τι γίνεται, να ξεπεράσουμε τα μεγάλα εμπόδια, ε, τα χωροταξικά, τα γεωγραφικά ποια είναι. Στο νότο οι Άλπεις, στο βορρά οι θάλασσες. Αυτά είναι τα έργα που πρέπει να γίνουν και τελικά να μπουν και διόδια για να προσελκύσεις και επενδυτές και ε, ιδιώτες επενδυτές που θέλουν να έχουν και κάποια απόδοση και κάποιο κέρδος. Όλα τα υπόλοιπα δεν λειτουργούν. Αυτό θα ε, ε, άρχιζε από το έργο ε, της σύραγγας του Μπρένερ. Προσπαθήσαμε να το κάνουμε στο παρελθόν με ευρωομόλογα και πάει λέγοντας ειδού ένα πολύ συγκεκριμένο έργο». Κοιτάξτε τι κάνει η Ελβετία. Το μεγάλο διάδρομα Γένοβα-Ροτερντάμ περνάει από δύο ε, μεγάλες σύραγγες Λόσπαξ στην Ελβετία και Γκοτάρδου που είναι με ιδιωτική επένδυση και πίπτει ράβδο στα διόδια. Και όταν περνάμε εμεί οι Ευρωπαίοι, πληρώνουμε βάζοντα το χέρι βαθιά στην τσέπη, θα μπορούσαμε λοιπόν στον Μπρένερ να κάνουμε το ίδιο. Τα ίδια ισχύουν για τη Σκανδιναβία και τη θάλασσα ε, για τις διασυμβέσεις. Ε, αυτά τα πράγματα είναι για μένα Connecting Europe Facility ή διευρωπαϊκά δίκτυα ε, μεταφορών στο μέλλον να τα χρηματοδοτούν οι χρήστες και ε, θα έχουμε τη δυνατότητα μετά στα διασυνοριακά που είναι πολύ σημαντικά ε, να περισσεύουν λεφτά. Και το ίδιο ισχύει για τον ορίζοντα 2020. Οπότε θα είχαμε πολύ μεγαλύτερο περιθώριο λιγμών για να χειριστούμε αυτά τα πράγματα. Ευχαριστώ. Θα ήθελα να θυμίσω ότι η ιδέα για ένα τέτοιο μεγάλο όγκο επενδύσεων προέρχεται βασικά από τα κράτη-μέλη. Γιατί καταπολέμηση τη ανεργίας, θυμάστε, αυτός ήταν ο λόγος. Διότι τώρα ε, διάφορα κράτη-μέλη έχουν ανεργία νέων 40 και 50% και η νεολαία τη δεν έχει ε, μέλλον. Και όταν σηκώνονται και φεύγουν οι νέοι, καταστρέφονται τα κράτη. Το ξέρουν και αυτοί. Και τα ξέρετε κι εσείς. Θα πρέπει λοιπόν να γίνει μια μεγάλη τέτοια ενέργεια για επενδύσεις για την καταπολέμηση της ανεργίας. Πουθενά όμως δεν έχω δει να γίνεται λόγος γι' αυτό. Ότι ναι, τα έργα θα πρέπει να είναι έτσι ώστε να δημιουργούν πολλές θέσεις εργασίας. Για να πάρουμε το δικό σας παράδειγμα. Ας πούμε βάλω μια μηχανή που να σκάβει μια σύραγγα κάτω από τη Βαλτική ή κάτω από τις Άλπεις μπορεί να είναι ωραίο αλλά δεν δημιουργεί θέσεις εργασίας. Ενώ εάν κάνουμε εξυγίανση ε, και ε, για τις υφιστάμενες υποδομές και στα κτίρια ε, δημιουργούνται θέσεις εργασίας και Ούτε κύχ δεν ακούμε γι' αυτό. Λοιπόν, τα κράτη που το ζητούν θα πρέπει να συμμετέχουν, όχι να πνίπτουν τα σχήρα του. Γι' αυτό πέρασε και έτσι γρήγορα από το Συμβούλιο. Δεν βάζουν ούτε σεντ, οπότε γιατί να είναι κατά. Παρά, μόνο κέρδο είναι όταν χτιστούν αυτά τα έργα. Και επίση η ανάλυση ότι η Ευρώπη θα πρέπει να ε, αυξάνεται ε, από κοινού. Το προσπαθούμε 20 χρόνια και να αναπτύσσεται με πάρα πολύ μικρή πρόοδο. Και ρώτησα τον μας πώς το βλέπει. Αν έρθουν ας πούμε αυτά τα 315 δις, θα έχουμε εμείς 100 εκατομμύρια έτσι ώστε το έτος 2016 να ε, ε, βάλουμε ε, σιδηρόδρομο μέχρι την πολιτιστική πρωτεύουσα της Ευρώπης. Μα μου είπαν με ξαναρωτήσατε και τώρα με ξαναρωτάτε. Ναι, σε ρωτάω. Γι' αυτό ρωτάω, διότι δεν με έχει δοθεί απάντηση θα μου δώσει απάντηση τώρα. Έχουμε ολόκληρη πολιτιστική πρωτεύουσα, το Πρέσλαο, χωρίς τρένο. Το 2016, αν δεν μπορούμε να έχουμε σιδηροδρομική σύνδεση, αλλά να κλείσουμε και αυτές που υπάρχουν, μία παραμονές Χριστουγέννων και μία μετά τα Χριστούγεννα, αυτό είναι αποτυχία για την Ευρωπαϊκή Ένωση και, και είναι και, και εκτεθειμένη. Και εκεί εμείς αποκλειόμαστε ότι καλούμεθα να πληρώσουμε, ε, ενώ την Επιτροπή Μεταφορών δεν έχουμε και λόγο. Και καθίστε στην άκρη μας, λένε θα τα κάνουμε εμείς. Δεν επιτρέπονται αυτά τα πράγματα, βεβαίως υπάρχουν εναλλακτικέ. Ο κύριος Μπέργκ έχει προτείνει μία από τον προπολογισμό του Κοινοβουλίου. Αν του περικόψουμε 1% τα χρηματοδοτούμε όλα. Οπότε δεν χρειάζεται το Connecting Euro. Αν έχουμε δυόμιση ε, από την Επιτροπή ε, Γεωργίας, ε, θα είχαμε πολλά λεφτά, αλλά εκεί θα εξαγριωθεί ο βασιλικός οίκος της Αγγλίας, γιατί παίρνει πολλά λεφτά για τη Γεωργία. Υπάρχουν λοιπόν λες λύσεις και λεφτά υπάρχουν, χωρίς να... προχωρήσουμε. και συμφωνούμε. Το είπα και στην διάσκεψη των Πρόεδρων. Στην Επιτροπή Μεταφορών συμφωνούμε και είμαστε όλοι υπέρ της συναπόφασης θέλουμε να δώσουμε ε, τις ιδέες μας και πρέπει να τα αλλάξουμε. Και η πολιτιστική πρωτεύουσα το 16 είναι το Βρόσλαφ Λοιπόν, δίνω το λόγο στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ο κύριος Βενιαμίν Άγγελ, Έγγελ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Angel είναι η σωστή προφορά. Άγγελος, όπως θέλετε, κύριε Πρόεδρε. Όπως θέλετε. Εντάξει, κύριε Άγγελε, έχετε το λόγο. Να ευχαριστήσω τους συνεισηγητές για την ταχύτητα με την οποία ετοίμασαν την έκθεσή τους να κάνω παρατηρήσεις σε πέντε τομεί για τον προπολογισμό, τις κατευθυντήριε για τις επενδύσεις, ε, την Επιτροπή Επενδύσεων, τον Διευλό και επειδή έρχομαι και από τη Γενική Διεύθυνση επειδή έρχομαι από τη συγκεκριμένη Γενική Διεύθυνση θα μιλήσω και για το Σύμφωνο Σταθερότητας και Να πω ότι έτσι όπως τα είπατε, είναι, φαίνεται, σας φάνηκε εύκολη απόφαση για τα κράτη-μέλη να πάρουν κονδύλια από το Connecting Group Facility και το Horizon 2020 όταν δεν έχουν διάθεση να συνεισφέρουν. Δεν είναι καθόλου έτσι τα πράγματα. Αν βλέπατε πώς πήγαν οι διαπραγματεύσεις στο Συμβούλιο και είχαμε δυσχερέστατες συζητήσεις με το Συμβούλιο και πολλά κράτη-μέλη που είχαν ακριβώ τι ίδιες ε, επιφυλάξεις που κι εσείς Γίνεται. Να πω ότι καταλήξαμε στα συμπεράσματα που όλοι γνωρίζετε. Ήταν το καλύτερο, ο καλύτερος δυνατός ε, ε, συνδυασμός. Τα κράτη-μέλη θέλουν να στηρίξουν το επενδυτικό πρόγραμμα. Ε, υπάρχουν ε, πολλά στο επίπεδο του Ταμείου που θέλουν να συμβάλλουν, αλλά το ίδιο και στο επίπεδο των επενδύσεων και στο επίπεδο των τραπεζών. Ε, την τελευταία εβδομάδα μόνο πέντε κράτη-μέλη μα έχουν ενημερώσει για τι εκπροθέσεις του και αν τις προσθέσουμε τις προθέσεις αυτές φτάνουμε μόνο τα 26 δις ευρώ. Ε, οπότε μην νομίζετε ότι τα κράτη-μέλη δεν θέλουν να συνεισφέρουν. Ίσα ίσα θέλουν να συνεισφέρουν προθυμότατα και εργάζονται εγκάρδια ε, προς αυτή την κατεύθυνση. Ως προς το δύσκολο σκέλος, δεν καταλαβαίνω ότι είναι και ευάλωτο για την, ε, ευαίσθητο για την Επιτροπή σας, ε, τις περικοπές του Connecting Europe που θα θελείτε. Ε, ανησυχεί πολύ η Ευρωπαϊκή Επιτροπή με την πρότασή σας να διαγραφούν τα άρθρα 18 και 19. Χρειαζόμαστε οπωσδήποτε να απελευθερώσουμε χώρο κάτω από την οροφή και γι' αυτό η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενδεικτικά έχει αναφέρει τις υποχρεώσεις από τις οποίες ε, σκοπεύει να κάνει περικοπές. Ότι θα πάρουμε δύο δις για το περιθώριο που αποκλειστικά όμως δεν μπορούμε να τα διαθέσουμε εκεί, το αναφέρατε πολύ από εσά. Αλλά υπάρχουν τρεις λόγοι για τους οποίους ανησυχούμε με την πρόταση αυτή του κοινοβουλίου για διαγραφή. Πρώτον, εάν δεν προβλέψουμε σαφή χρηματοδότηση εκ των προτέρων, οι αιτήσει συζητήσει για τον προπολογισμό θα γίνουν ακόμη πιο χαοτικέ από ό,τι είναι ήδη. Θα μπορούσε βεβαίω κανεί να ισχυριστεί ότι από την σκοπιά του Κοινοβουλίου είναι ήδη δύσκολα τα πράγματα, αλλά υπάρχουν και άλλοι δύο λόγοι. Ο ένα είναι ότι χρειάζεται προβλεψιμότητα στον τρόπο με τον οποίο διαχειριζόμαστε τα προγράμματά μα και αν για βασικούς τομείς δαπανών υπάρχει αβεβαιότητα κάθε χρόνο σε επί σειρά ετών για το πόσα μπορούμε να δαπανίσουμε, θα γίνει άκρος δύσκολο να προγραμματίσουμε τη δαπάνες. Υπάρχει ένα σωρό από, υπάρχουν ένα σωρό τομείς όπου οι δαπάνες ξεκινούν σε πολιτή βάση, όπως με την έρευνα. Τρίτον, σε ένα τοπίο όπου ήδη έχουμε την, τα 26 δις ε, ευρώ σε backlog και τα οποία δεν πληρώνονται, το να πληρώσουμε το να, μια εγγύηση 16 δις που δεν θα μπορούμε να δικαιολογήσουμε ή να αιτιολογήσουμε στους διάφορους οργανισμούς, πώς ακριβώς χρηματοδοτήθηκαν, αυτό θα κάνει την πιστοληπτική ικανότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης πολύ αμφίβολη. Θα κινδυνεύσει πολύ. Ξέρω λοιπόν ότι α, η ΕΤΕ πρέπει να προστατεύσει τον τριπλό της Α και ιδίως από τους οίκους ε, αξιολόγησης. Οπότε ε, πραγματικά ε, θα πρέπει να συστήσω στα μέλη του να σκεφτούν πολύ καλά το πώς μας απασχολεί αυτή η πως την οπτική μας ικανότητα για να είναι τα ομόλογα επιλέξιμα πρέπει να έχει κανείς τριπλό α τουλάχιστον από δύο από τους τρεις μεγάλους οίκους αξιολόγησης. Ένας και μόνο να υποβαθμίσει την τράπεζα θα είναι φοβερά αρνητικό αντίκτυπο για την πρόσβαση στην αγορά, από την αγορά τη ΕΕ. Το λέμε λοιπόν για όσου από εσά θεωρούν ότι δεν μπορούμε να αφήσουμε άδειο το κουτί της χρηματοδότησης. Εάν δεν σας αρέσει κάτι στο πρόγραμμα χρηματοδότησης, να μας δώσετε μια πλήρως διαφρωμένη εναλλακτική πρόταση. Αλλά δεν μπορείτε να τα αφήσετε ανοιχτό, χωρίς να εκτεθούμε σε πολύ σοβαρό κίνδυνο. Σε ό,τι αφορά τον προπολογισμό, να τονίσω επίσης ότι παρά το γεγονό ότι παίρνουμε από υποχρεώσει ε, σημαντικών προγραμμάτων, σημαντικά και για την ίδια την Επιτροπή άλλωστε, δεν το κάνουμε αυτό με την προσπάθεια να κάνουμε λιγότερα, κάνουμε ό,τι μπορούμε ε, και μάλιστα θα κάνουμε και περισσότερα στους ευλογοτομείς. Όταν ε, παίρνει κανείς ε, χρήματα από τις δωρεές υπάρχει μόχλευση 1 έως 3 το πολύ. Και εάν κανείς τα τοποθετήσει ε, προβλεπόμενες προβλεπόμενε επενδύσει με πολλαπλασιαστή 15, με μόχλευση 15, τότε η Επιτροπή μπορεί να υποσχεθεί ότι θα υπάρξουν πολύ περισσότερε δράσει για τι μεταφορέ από ό,τι αρχικά γινόταν. Δεύτερο τομέα, οι κατευθυντήριε γραμμέ για τι επενδύσει. Είναι πολύ σημαντικό για μα τα εργαλεία να είναι ευέλικτα επανειλημμένω έχουμε δει πολύ καλά εργαλεία να ε, κατατρέφονται λόγω του περίπλοκου χαρακτήρα τη χρήση του. Όπω τα ε, ομόλογα ρήγων. Ήταν ένα εργαλείο του οποίου η λειτουργία δεν διαφέρει πάρα πολύ από αυτό που τώρα σχεδιάζουμε. Θα μπορούσε κανεί να έχει ένα φανταστικό έργο σήμερα στην Πορτογαλία και να μην μπορέσει να το χρηματοδοτήσει. Γιατί μια από τι προποθέσει είναι ότι πρέπει να είναι διακρατικό. Οπότε ε, θα πρέπει θα πρέπει να αποφύγουμε τις δυσκολίες ε, με τις κατευθυντήρες για τις επενδύσεις, ώστε να είναι ευέλικτη στη χρήση, γιατί ένας ελβετικός σουγιάς μας χρειάζεται, ε, για να μπορούμε να προκαλέσουμε τις επενδύσεις που θέλουμε, χωρίς γεωγραφικό εντοπισμό, ούτε τομεακό εντοπισμό. Θέλουμε πλήρη ελευθερία. Ταυτόχρονα θα πρέπει να συμφωνήσουμε όλοι ότι δεν θα υπάρχει υπέρμετρη έκθεση στο κείμενο για έναν συγκεκριμένο τομέα ή για ε, μια συγκεκριμένη γεωγραφική περιοχή. Αυτό θα πρέπει να συμπεριληφθεί ξεκάθαρα στι γραμμέ για τι επενδύσει. Είναι σαφή πρόθεση τη Επιτροπή. Τρίτη παρατηρήση. Η Επιτροπή Επενδύσεων. Η Επιτροπή αυτή είναι ακρογωνιαίο λίθο τη πρόταση. Πρέπει να σα θυμίσω ότι δεν συζητούμε εδώ μια νέα εκδοχή των διευθυντικών ταμείων ή ένα νέο πρόγραμμα για δωρεές. Η πρόθεση του προγράμματος Juncker δεν είναι να πολλαπλασιαστούν οι δημόσιες επενδύσεις. Η πρόθεση του προγράμματος Juncker είναι να χρησιμοποιήσουμε όσο το δυνατόν λιγότερο δημόσιο χρήμα για να προσελκύσουμε όσο το δυνατόν περισσότερο ιδιωτικό χρήμα για να χρηματοδοτήσουμε τι επενδύσεις μας. Για το σκοπό αυτό χρειαζόμαστε οπωσδήποτε βεβαιότητα ότι οι επενδύσει επιλέγονται από ένοξη, ανεξάρτητους εμπειρογνώμονες της αγοράς χωρίς καμία πολιτική διάσταση στην διαδικασία. Αν αρχίσουμε να δίνουμε πολιτικό χαρακτήρα στη διαδικασία, μπορεί να ε, βάλουμε τρικλοποδιά στον εαυτό μα και να ε, επηρεάσουμε το δομή των συζητήσεων, μπορεί να είναι ενδιαφέρουσε, αλλά σίγουρα δεν θα πείσουμε του επενδυτέ, οι οποίοι ε, ενδιαφέρονται για την λογική τη επιλογή των έργων. 80% των κονδυλίων του προγραμματό θα έρθουν υποτίθεται από τον ιδιωτικό τομέα. Ο μόνος τρόπο να το βεβαιώσουμε αυτό είναι να γίνει με τρόπο έμπροστο και πολύ καλά προετοιμασμένο χωρί να υπάρξει καμία εξωτερική παρέμβαση. Μην θεωρείτε λοιπόν ότι το Κοινοβούλιο ε, θα πρέπει να συμμετέχει στην εργασία τη Επιτροπή Επενδυτών, ούτε η ΕΤΕ θα πρέπει να συμμετέχει, ούτε ε, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η ε, Επιτροπή Επενδύσεων θα πρέπει να υλοποιήσει με τρόπο γράφειο κρατικό τι στρατηγικέ γραμμέ που θα έχουν αποφασιστεί βάσει των αρχών που θα καταγράψουν και θα κατοχυρώσουν τον κανονισμό οι συνομοθέτες. Τέταρτη παρατήρηση για την διαβλό. Την... Έχω δει στο σχέδιο έκθεση ε, να υπάρχουν κάποιε δυσκολίε κατανόηση και καλά τα εντόπισαν οι συνεισηγητέ, ε, διότι έχει μπερδέψει πολλού. Δεν έχει καμία σχέση με το πρόγραμμα και ο διαβλός. Μάλλον με το έψη αυτό καθεαυτό δεν έχει σχέση. Διότι το πρόγραμμα το έργο που θα βρίσκεται στον διάβλο προετοιμασία δεν, δεν καθορίζει το, η θέση του αυτή το κατά πόσο θα χρηματοδοτηθεί από το ΕΦΣΙ ή από την ΕΤΕ. Απλώ θέλουμε να υπάρχει ένα ξεκάθαρο ιστότοπο με τι επενδυτικέ ευκαιρίε στην Ευρώπη, όπου τα έργα συγκεκριμένων διαστάσεων και μεγέθου που θα είναι συμβατά με την πολιτική αυτή, θα μπορούν να ε, αποτελέσουν πόλο έλξη για του ίδιου του επενδυτέ. Θα πρέπει η διαδικασία να είναι διαφάνεια και παρουσίαση των έργων, αλλά με τι επενδυτικέ ευκαιρίε, όπου κάποιε φορέ θα θέλουμε να αποφύγουμε και το παραμικρό λεπτό του ευρώ από δημόσια κονδύλια ή δημόσιο προπολογισμό θα είναι καινοτόμο το εργαλείο αυτό. Είναι μια πολύ καινοτόμα προσέγγιση, γιατί δεν υπάρχει προηγούμενο πουθενά στον κόσμο και είναι ιδιαίτερη σημασία και ιδιαίτερα ελκυστικό για τα μικρά κράτη-μέλη. Αυτά που κατά τρόπο φυσικό δεν είναι έλξη για του επενδυτέ. Αν είναι κανεί στη Γαλλία ή τη Γερμανία, βεβαίω υπάρχει περιθώριο για επενδύσει. Εάν είναι κανεί όμω στι χώρε τη Βαλτική ή στι νότιε ε, ακτέ τη Ευρώπη, τα πράγματα είναι ίσω πολύ πιο περίπλοκα για του επενδυτέ. Δεν έχουν τι πληροφορίε που θέλανε. Οι επενδυτέ ενώ τώρα θα έχουν πρόσβαση σε έναν ενιαίο ιστότοπο με έναν τρόπο πολύ εύληπτο. Όμω κανεί δεν χρειάζεται να αγωνιστεί για το θέμα αυτό, τι θα είναι το pipeline αυτό ο διάβλο και τι ε, θα περιλαμβάνει. Ό,τι θα αποστέλλεται και θα, ε, έχει, τις πληρεί τι προποθέσει θα συμπεριλαμβάνεται στο pipeline χωρί να έχει σχέση με τα υπάρχοντα και τρέχοντα έργα. Ε, και μετά για το Σύμφωνο Σταθερότητα και Ανάπτυξη. Είδαμε ότι η Επιτροπή σα, μαζί με τι υπόλοιπε κοινοβουλευτικέ επιτροπέ, κάνει την πρόταση να το αξιοποιήσουμε με ένα συγκεκριμένο τρόπο το σύμφωνο. Εδώ πρέπει να πω το εξή. Θα πρέπει να σας βάλω λίγο πάγο. Διότι και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή Στοματοφύλακας των Συνθηκών γνωρίζει ότι η νομική βάση για τον κανονισμό αυτό κατά πρώτον δεν επιτρέπει καθόλου την τροποποίηση του Συμφώνου Θεώτος και Ανάπτυξης. Υπάρχει νομική βάση για την βιομηχανία την έρευνα εδώ, αλλά πέραν αυτών το Σύμφωνο σταθερότητα και ανάπτυξη είναι κανονισμό του Συμβουλίου. Και είναι κανονισμό του Συμβουλίου γιατί η συνθήκη έχει συνταχθεί κατά αυτόν τον τρόπο και θα καταλαβαίνετε ότι είναι πολύ δύσκολο να το πω διαφορετικά. Δεν μπορεί το Κοινοβούλιο να τροπολογήσει κανονισμό του Συμβουλίου με ένα κείμενο συναπόφαση πέραν του θέματος τη νομική βάσης, έτσι και Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν μπορείτε να κάνετε προτάσεις Όμω οι προτάσεις σας καλό θα είναι να γίνουν με ψηφίσματα λόγου χάρη. Αυτό θα ήταν το καταλληλότερο εργαλείο για να προχωρήσετε. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ο Ντομινί Κρικέ, ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Προσπαθήσω να είμαι σύντομος ε, και συνοπτικός. Σε αδρές γραμμές υπάρχουν δύο δέσμες, δύο πτυχές. Ρύθμιση του μηχανισμού αφενός και προέλευση των κονδυλίων για το Ταμείο Εγγύησης αφετέρου. Σε ό,τι αφορά το μηχανισμό, δύο θέσεις ακούσαμε ότι υπάρχουν. Τη μία την υπερασπίζεται η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και την άλλη πράσινη, για παράδειγμα, οι σοσιαλιστές. Δηλαδή, από τη μια πλευρά ότι δεν πρέπει να περιπλέξουμε τα πράγματα αντίθετα να τα απλουστεύουμε και να μην παρεμβαίνουμε τόσο πολύ στη λειτουργία του συστήματος γιατί η άγρα επενδυτών είναι σαν να κυνηγάμε ε, το θύραμα αλλά πρέπει να είμαστε σιωπηλοί και ίσοι για να μην φύγει. Ε, επομένως δεν θα πρέπει να έχουμε ε, πάρα πολύ επεμβατικό τρόπο να πετύχουμε τους στόχους μας. να μην περιπλέξουμε τη λειτουργία του συστήματος. Θα προσπαθήσουμε να βρούμε το μέτρο μαζί με την Ινές. Το δεύτερο είναι η προέλευση των ε, χρημάτων. Εδώ είναι το ζήτημα, το κεντρικό. Νομίζω ότι οι περισσότεροι όσοι πήραν το λόγο είπαν ότι δεν δέχονται τα άρθρα 18 και 19. Δηλαδή δεν θα, δια... θα δεχτούμε να μας αδειάσουν τις ε, τσέπες και όχι μόνο τις τσέπες αλλά και το κεφάλι. Ιδίως ε, σε ό,τι αφορά ένα μηχανισμό που αποτέλεσε αντικείμενο διαπραγματεύσεων πολλά χρόνια και δεν θα πάμε να του στερήσουμε τη χρηματοδότηση αυτού του μηχανισμού. Αυτό πρέπει να το καταλάβει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Τώρα άκουσα αντιθέτω ότι υπήρχαν προτάσεις να πάμε πιο μακριά από αυτό που προτείνουν οι δύο εισηγητές. Ναι, το κατανοώ, αλλά πρέπει και να το συζητήσουμε. Υπάρχουν ε, συγκεκριμένα εμπόδια ενδεχομένως για να προχωρήσουμε πιο πέρα. Ολοκληρώνοντα να πω δύο λόγια για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, τον εκπρόσωπό τη τον άκουσα όπω πάντα με πολύ μεγάλη προσοχή και θα έλεγα και με ιδιαίτερη χάρα διότι βλέπω ότι υπάρχουν ε, κάποια κοινά σημεία, συμφωνούμε σε ό,τι αφορά τι δυσκολίε για παράδειγμα. Εμεί στην έκθεσή μα εμείς δεν σκεφτήκαμε κάτι διαφορετικό για αυτό το pipeline, αυτή τη δεξαμενή έργων. Βέβαια πρέπει να σας ομολογήσω μόνο ότι δεν έχει καμία σχέση με το Ταμείο Στατικών Επενδύσεων. Τότε τι δουλειά έχει σε αυτό το κείμενο. Έτσι μας είπατε ότι δεν έχει καμία σχέση με το Ταμείο Στατικών Επενδύσεων. Πού φύτρωσε λοιπόν, πού ξεφύτρωσε μέσα στο κείμενο αυτή η δεξαμενή, αυτό το pipeline. Δεν πρέπει να μας βρείτε μια καλύτερη εξήγηση. Άρθρο 18 και 19, καμία σχέση ε, πάλι με το Ταμείο Στατικών Επενδύσεων έχουν να κάνουν τον προπολογισμό. Βέβαια το θέμα του Ταμείου Εγγύσεων είναι πολύ σημαντικό ζήτημα. Συμφωνώ με αυτά που είπατε για το Σύμφωνο Σταθερότητα. Θα έπρεπε να το συζητήσουμε μεταξύ μα. Είναι ένα μήνυμα που εμεί θέλουμε να εκπέμψουμε τον ένα τον άλλο τρόπο, ότι δεν θα πρέπει δηλαδή ε, με ένα τέτοιο ε, σύστημα, σε ένα τέτοιο μηχανισμό, να τιμωρήσουμε τις χώρες που βρίσκονται σε δυσχερή θέση. Το αντίθετο θα πρέπει να κάνουμε. Δεν θα πρέπει να αφήσουμε να πεθάνουν από την πίνα αυτοί που πεινάνε. Πρέπει να είμαστε λίγο πιο ισορροπημένοι στην προσέγγισή μας. Καταλαβαίνω επίσης πολύ καλά την ανησυχία που εξέφρασε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε ό,τι αφορά τη σταθερότητα της ΕΤΕ, την βαθμολόγηση, την αξιολόγησή της δηλαδή, το rating κτλ. Τώρα, σε ό,τι αφορά τη δική σας παρέμβαση για τον προπολογισμό, Άκουσα πάρα πολύ προσεκτικά ε, και με χαροποίησε ότι δεν υπάρχει κανένα επιχείρημα. Εγώ περίμενα να μπορέσετε να μας πείσετε, αλλά τουλάχιστον εμένα δεν θα με πείσετε. Λέτε, η καλύτερη θέση είναι αυτή της Κομισιόν. Έτσι ξεκινάτε και βέβαια πράγματι είναι βάση για την όλη συζήτηση. Αν μας εξηγήσετε όμως και αν μας πείτε ότι δεν θα είναι και πολυβολικό να κάνουμε κάτι διαφορετικό γιατί θα είναι το Λίπρο και συζητήσει για την κατάρτιση του υπερπολισμού. Τα τελευταία χρόνια θέλω να σα πω ότι έχω λάβει μέρο και στη συζήτηση για τον υπερπολισμό και σε πολλού τρομερεί και πάντα ήταν πολύπλοκη όλη η διαδικασία. Το να υπάρξει λοιπόν ένα επιπλέον κεφάλαιο για ένα δι ή ένα μισή δι δεν θα περιπλέξει περισσότερο τα πράγματα. Δηλαδή μπροστοβαρή εκταμίευσή του, λιγότερο τα επόμενα χρόνια, περισσότερο τα πρώτα. Εγώ θέλω να επιστήσω την προσοχή των συναδέλφων μου, αλλά και της Κομισιόν, στο γεγονό ότι ναι, θα ακούσουμε το επιχείρημα. Δεν μπορούμε να υποβαθμίσουμε την ε, αξιοπιστία του μηχανισμού, γιατί αυτό το Ταμείο Εγγύσεων δεν είναι εγγύηση. Αν διαβάσετε όμως προσεκτικά την έκθεση, θα καταλάβετε ότι είναι εγγύηση, γιατί τελικά αυτά τα δύο ταμεία είναι η βάση. αυτά στηρίζεται, σε αυτό το μηχανισμό που αναφέρεται. Ε, πρέπει να πω επίσης ότι η πρόταση που σας ε, κάνουμε είναι υπάρχουν ε, μη διατεθήσεις πιστώσεις. Αυτές οι μη διατεθήσεις πιστώσεις στον προπολογισμό θέλουμε να διατεθούν κατά προτεραιότητα και νομίζω ότι είναι καλύτερο να γίνει αυτό. Και τώρα μας λέτε ότι έχουμε 26 δις ανεξόφλητους λογαριασμούς στον χρόνο ε, και κάθε χρόνο σωρεύονται ακόμη περισσότεροι. καταλαβαίνετε ε, ότι υπάρχουν και πολλά ποσά που γυρίζουν πίσω στα κρατημέλη που δεν έχουν όμως καταβάλει ε, αυτά που όφυλαν. Μας ανησυχεί πάρα πολύ το θέμα των εξόφυτων λογαριασμών. Όλους τους ευρωβουλευτές. Δεν μπορούμε όμως να ανεχθούμε από αυτές τις συνθήκες να έχουμε εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ που θα επιστρέφονται κάθε χρόνο στα κρατημέλη. Μην μας λέτε λοιπόν ότι το χάος του προβληματισμού ή ανεξόφλοι λογαριασμοί είναι επιχειρήματα για να μην πάμε σε μια χρήση αυτών των μη πιστώσεων στο Ταμείο Εγγύησης. Και υπάρχει και ένα σκάνδαλο, τα κράτη-μέλη. Ένα μέρος των προστήμων τα διατήρησαν, τα βάλανε στις τσέπες, αν θέλετε, στα, στα ταμεία τους, χωρίς να έχουν εξοφλήσει τους οργανισμούς. Δεν μπορούμε να τα ε, δεχόμαστε αυτά από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Εγώ νομίζω ότι μπορούμε να διαχειριστούμε τις μη διατηρήσεις πιστώσεις με σωστό τρόπο. Μας λέτε επίσης, με αυτό το μηχανισμό θα κάνουμε περισσότερα. Με αυτό το Ταμείο δηλαδή, Επίσης για τον τομέα των μεταφορών, την έρευνα για παράδειγμα. Είχα όμως την τιμή και τη χαρά να συμμετάσχω στον τομερή διάλογο για το Connecting Europe Facility και πρέπει να σας πω ότι τα κράτη-μέλη δεν ήθελαν να ακούσουν για κανένα χρηματοδοτικό μέσο που μας λέτε ότι μπορεί να είναι καλύτερο. Και δεν ξέρω εγώ με ποια μόχλευση για να φτάσουμε σε ένα τεράστιο ποσό από τα κράτη-μέλη. Μια πολιτική που ποτέ δεν την υποστήριξαν, θέλουν να τη χρηματοδοτήσουν με, με τα ευρωπαϊκά ε, κονδύλια, τα κράτη-μέλη. Σίγουρα είναι πολιτικό το σχέδιο Γιούγκερ ε, υπό την αγίδα του, αλλά δεν πιστεύω ότι το έχει πιστέψει. Ε, πρέπει να δούμε τελικά πόσο σοβαροί είμαστε στην κατάσταση προβλησμού, πώς μπορούμε να αξιοποιήσουμε τα κονδύλια με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Είχαμε δάνεια, είχαμε τις επιχορηγήσεις και τώρα ακολουθούν μια θεωρητική γλώσσα. Εγώ θα έλεγα ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή καλό θα ήταν να επανέλθει στην αρχική της τοποθέτηση που ηθικά ήταν υποστηρίξιμη και ήταν και ορθόδοξες από πλευράς δημοσιονομικής. Ενώ δεν ισχύει το ίδιο με αυτές τις προτάσεις. Υπάρχουν μη διατεθήσεις πιστώσει ας τις διαθέσουμε για αυτό το μηχανισμό και να διατηρήσουμε τελικά και κάποιους πόρους για αυτό το ταμείο, για να έχουμε αυτή την εγγύηση, γιατί μα είπατε ότι υπάρχει κάποια αλλίωση των ε, πολιτικών της Ένωσης. Αυτό γίνεται λόγω του Συμβουλίου, όχι λόγω της επιχειρηματολογίας του Κοινοβουλίου. Αυτά έχω να πω προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Νομίζω ότι τα επιχειρήματα που τα ακούσαμε και θα τα ξανακούσουμε και στους τριμερείς έλεγχους δεν πρόκειται να πείσουν το Κοινοβούλιο. Και υπενθυμίζω ότι καλό θα ήταν να φτάσουμε σε μια κοινή θέση αν θέλουμε αυτός ο μηχανισμός τελικά να λειτουργήσει, να ευδοκιμήσει. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ η κυρία Γιάλα Σέντερ. Έχει το λόγο. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Πρώτο. Επιβεβαιώνω τα όσα είπε ο κύριος Ρικέ, συνάδελφος. Καταρχήν θα πρέπει να φροντίσουμε να είναι αξιόπιστος ο ευρωπαϊκός προπολογισμός για να μπορεί να δώσει εγγύηση να σταματήσει αυτό το παζάρι και το παιχνιδάκι των κρατών μελών, να έχουμε ένα δις ε, κάθε χρόνο ε, που αρνούνται να, να πληρώσουν. Εν πάση περιπτώσει κάθε χρόνο έχουμε περίμερες και ανεξόφλητες ε, πιστώσεις. Θέλω να διευκρινίσω μερικά πράγματα. Σε σχέση με τα έργα που αν συμμετείχαν ή όχι και στη διαβούλευση οι αρχέ τη τροπική αυτοδιοίκηση. Δεν μιλώ τώρα για τη συζήτηση για το Ταμείο. Απλώ θέλω να καθησυχάσω όλου του συναδέλφου που δεν έχουν παρακολουθήσει όλη αυτή τη μακρά πορεία ε, της ε, Connecting Europe. Στο άρθρο 5α ακριβώ. αναφερόμαστε σε αυτό. Ε, τα προγράμματα και τα έργα του σχεδίου Juncker έχουν σχέση με τους δύο μεγάλους κανονισμούς του Connecting Europe και εκεί μένουν και τα μικρά διευρωπαϊκά δίκτυα, τα διασυνοριακά. Ε, έχω και ίδιο <laughs> συμφέρον εγώ. Επίσης γίνεται λόγος για ε, όλες τις αρχές τοπικής αυτοδιοίκησης που θα ήθελα να μας δώσουν την άποψή τους. Καλέσαμε. Να μην ανησυχεί κυρία Ντελή γιατί άμα εγκριθεί το 5α εκεί προβλέπεται όλη αυτή η συζήτηση και ε, έχουμε συμπεριλάβει όλες τις ανησυχίες και τα μελήματα και για τα τοπικά διασυνοριακά δικτύα ακόμα και όλες τις δυνατότητες να προχωρήσουμε ακόμα παραπέρα. Όλα αυτά στα πλαίσια των αρχών και των αξιών που διέπουν και αφορούν την Ευρώπη, από τις οποίες εμφορείται μόνο η Ευρώπη. Έχετε δίκιο. Δεν είναι μόνο επιδοτήσεις, υπάρχουν και άλλα χρηματοδοτικά μέσα. Δεν είναι κάτι που έχουμε εφεύρει τώρα. Τα ομόλογα έργου υπάρχουν ήδη ως δυνατότητα και από τους συνδέοντας στην Ευρώπη. Το θέμα είναι ότι τα κράτη-μέλη δεν επίστευαν πάρα πολύ σε αυτά και χρειάστηκε να πιέσουμε για να υπάρχει ένα, κλάσμα για να μπορέσουμε να μοχλεύσουμε με ιδιωτικές επενδύσεις πέρα από τις δημόσιες. Ο, ο κύριος Πίπερ βλέπω να επιμένει πέρα από τις διάφορες δυνατότητες διεύρυνσης του προϋπολογισμού, όπως είπε και ο κύριος Ρικέ, και ως έσχατη λύση να μπορέσουμε να επανέλθουμε στον τίτλο 1α, είμαι απολύτω αντίθετη με το να δημιουργήσουμε και νέα σύγκρουση και νέα σύγχυση και νέα ε, ασάφεια και στο ένα, προσπαθώντας να βάλουμε και το ένα β Έτσι κι το Συμβούλιο από την αρχή είπε δεν βάζω ούτε δεκάρα. Και η κυρία Μέρκελ από την αρχή, ε, ε, από το κοινό ταμείο. Δεν μπορούμε όμως τώρα να πάρουμε λεφτά από τους γεωργούς. Δηλαδή, οι δικοί μου ε, ε, έχουν ε, πρόβλημα από το εμπάργκο της Ρωσίας πρώτη χρονιά, τώρα πάει, τρέχει δεύτερη χρονιά και ποιος θα πάει να πει στους γεωργούς του ότι μας δώσαν 10 δις ας πούμε για τη διευκόλυνση συνδέοντας την Ευρώπη που ακόμα πρέπει να ε, τους ευχαριστούμε για χώρες που δεν είμαστε στη συνοχή για να βούμε στον διαγωνισμό, δεν θα πούμε τώρα ότι θα σας καβάρουμε το χέρι στην τσέπη στο 1β. Κύριε Πίπερ. καταλαβαίνω την πρόθεσή σας, αλλά καμιά φορά αναρωτιέμαι ε, αν θέλετε να πετύχει να αποτύχει το σχέδιο Juncker, πού το πάτε. Και να επιμένετε για το 1β, να πάτε να εξηγήσετε στους γεωργούς που είναι ήδη σε πάρα πολύ δίνη θέση και μετά στις περιφέρειες της χώρας συνοχής, πολλές φορές είναι γείτονέ σα, τι θα κάνουν και από πού θα ε, τους αφαιρέσετε αυτά τα κονδύλια. Γιατί τουλάχιστον ο κύριος Δικέ και εγώ μαζί με τους συναδέλφους του προϋπολογισμού έχουμε βρει ε, περιοχές, ας πούμε, κονδύλια από τον προϋπολογισμό πιστώσεις που δεν φύγουν αυτά που ανεφέραμε και ε, ακόμα και το ΣΕΦ και το ορίζον 2020 έχουμε δυνατότητες να τα βρούμε απαλού Να πω τώρα για τον κύριο Έντζελ Άγχελ, πώς σας λένε, εν πάση περιπτώσει. Θέλω να ρωτήσω από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή το εξή. Δεν συνηθίζουμε να συζητάμε ε, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή από τη Γενική Διεύθυνση ε, οικονομικών συζητάμε με τη Γενική Διεύθυνση Μεταφορών. Καλό θα ήταν ένα συντονισμό μεταξύ σα. Γιατί ε, μα λέτε ότι αν μπούμε στην γνωστή φόρμουλα του ετησίου προπολογισμού και των ε, ομολόγων έργου, αυτό θα σημάνει προβλήματα στην διασυνοριακότητα. Μα μπορούν να είναι και διμερεί τα ομόλογα έργου, μπορεί να είναι και μονοεθνή. Το σχέδιο Κάστορ που δεν ήταν το μεταφορών, ευτυχώ γιατί θα με είχαν ζώσει τα φίδια αλλά υπάρχουν προγράμματα εθνικά που ακριβώς ε, έχουν ε, συγχρηματοδότηση, ΣΔΙΤ και τα λοιπά. Δεν ευδοκίμησαν. Δυστυχώς όλα αυτά τα κριτήρια που μας λέτε δεν είναι εγγύηση για να λειτουργεί σωστά. Και σε ό,τι αφορά τους ανεξόφλητους λογαριασμούς, πολύ ωραία τα είπε ο κύριος Ρικέ. Στις ΗΠΑ Πολιτείες τι γίνεται. Με την κυβέρνηση Ομπάμα βλέπετε κάθε χρόνο το στριμώχνουν. και βέβαια δεν πιστεύονται, εμπιστεύονται, ναι. Δεν, δεν είναι, ε, βλέπετε, εμπόδιο ή ανεξόφλητοι λογαριασμοί όταν είναι ελκυστικό ένα έργο έρχονται οι επενδυτέ. Ε, δεν σημαίνει ότι έχουν γυρίσει την πλάτη στον κύριο Ομπάμα επειδή κάθε χρόνο δυσκολεύεται να πληρώσει τους υπαλλήλου του στο τέλο του χρόνου. Υπάρχουν δυνατότητε να δοθούν εγγυήσει με καλύτερο τρόπο και όχι ε, να παίρνουμε από τη μία τσέπη για να τα βάζουμε στην άλλη κάθε χρόνο. Υπάρχει ένα σχέδιο Juncker ήδη για τις υποδομές, αλλά θέλουμε διεύρυνση του ΣΕΦ, που τα είχε όλα, και χρηματοδοτικά μέσα, και έργα, και ελκυστικά και λιγότερο ελκυστικά, επιδοτήσεις, προσέγγισης, ΔΙΤ, ιδιωτικό τομέα, δημόσιο, τα πάντα και όλοι τα είχαν εγκρίνει, συμβούλιο, οι πάντες, τα κράτη-μέλη, περιφέρειες, η βιομηχανία, όλοι. Ε τώρα μην μας ξυλώνετε αυτό το μέσο που φτύσαμε αίμα να το φτιάξουμε και βοηθήστε μας, Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Βοηθήστε μας, γιατί και το Συμβούλιο τραβάει τη δική του γραμμή, για να έχουμε ένα σχέδιο Juncker και βοηθήστε μας ε, να μπορέσει ακόμα περισσότερο να υποστηρίξει στην Ευρώπη τις επενδύσεις και την ανάπτυξη. Εμείς μπορούμε να τους δώσουμε και να σας δώσουμε μια σειρά απολύσεις και θα πρέπει να μας βοηθήσετε αντί να μας στέλνει σημειώματα ο κύριος Κατάινεν που δεν βοηθάνε καθόλου την υπόθεση, ε, βοηθήστε μας να προχωρήσουμε, να τα βρούμε με το Συμβούλιο. Από τα 28 κράτη-μέλη, μόνο 5 έχουν εγγραφεί. Η δική μου χώρα, η Ισπανία, δεν μπορεί να δώσει δεκάρα ε, χωρίς να του ανάψουν όλα τα, καμπανάκια, ε, τα λαμπάκια και να χτυπήσουν όλα τα καμπανάκια του συμφώνου σταθερότητας πώς θα μας βοηθήσετε. Η ανακοίνωση του κυρίου Μοσκοβισή θα δούμε. Μπορεί να μας ανοίξει μια πόρτα και θα πρέπει να βοηθήσετε αυτά τα κράτη-μέλη, εσείς από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, να ε, δείξουν μεγαλύτερη προθυμία για το σχέδιο Γιούνκερ. Ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, η πρώτη εξέταση των τροπολογιών 26 Μαρτίου. Βέβαια μόνο στα αγγλικά είναι οι τροπολογίες. Η δεύτερη με μετάφραση όλων των τροπολογιών στις 13 Απριλίου πριν την ψηφοφορία. Δηλαδή 13 Απριλίου ψηφίζουμε και προηγουμένως έχουμε όλες τις τροπολογίες μεταφρασμένες. 25 Μαρτίου θα έχουμε την αγγλική μετάφραση online. Α, προθεσμία κατάσταση τροπολογιών και για τις δύο γνωμοδοτήσεις 19 Μαρτίου 2015, 12 το μεσημέρι. Ορίστε. Κάτι λέει ο κύριος Παντανκάμπ. Τώρα αυτή τη βδομάδα είναι, ναι. Είναι πολλά τα λεφτά, 315 δις. Μπορεί να είναι και λιγότερος ο χρόνος. 11 χρόνια είμαι στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ποτέ δεν έχω δει τέτοιο έργο και τόσο γρήγορα. Και ρωτάω την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Τι σας έχει πιάσει, γιατί βιάζεστε, 315 δισεκατομμύρια θα πρέπει να κοιτάμε σε λεπτομέρεια. Καλύτερα να χρειαστούμε μια εβδομάδα και ένα μήνα παραπάνω ή τώρα να περάσει οπωσδήποτε για τον Ιούνιο γιατί το έχουν εξαγγείλει. Πρέπει να έχει κάτι μέσα για να καταπολεμήσει την ανεργία, να σταματήσει την κλιματική αλλαγή και να φέρει πιο κοντά την Ευρώπη. Ε, τώρα το έχουν αποφασίσει, αυτά είναι, αυτές είναι οι ημερομηνίε με κάθε ταπεινότητα εγώ σας τις ανακοίνωσα. Ε, vote, also, η ψηφοφορία στην Επιτροπή μας είναι στις 14 Απριλίου, στη δε ολομέλεια, στη δεύτερη ολομέλεια του Ιουνίου του 2015. Εντάξει. Gut. Dann... Προχωράμε. Ενημέρωση σχετικά με τους τριμερείς διαλόγους και κλεισμένο των θυρών είναι για το σιδηροδρομικό πακέτο. Παρακαλώ να αποχωρήσουν όσοι δεν δικαιούνται να παρευρίσκονται στην και των θυρών συνεδρίαση. Βεβαίω όλοι οι βουλευτέ μπορούν να παραμείνουν.